να μην ήμουν πάντα ένας μετριοπαθής, αλλά πάντα προσπάθησα να προασπίσω την, το σωστό και τους ψηφοφόρους μου. Γιατί πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι κάτι που αξίζει να πολεμήσουμε για την ειρήνη και την κοινότητα. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι αυτή είναι η βασική ελπίδα για την οποία πρέπει να δουλέψουμε. Ευχαριστώ. Τζόφολη, δύο λεπτά για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Καλύτερα με το μικρόφωνο, κύριε συνάδελφε. Δεν υπάρχει μικρόφωνο, κύριε Τζόφολη. Συνεχίζετε να μην έχετε μικρόφωνο. Με ακούτε τώρα. Η ο κανονισμός που υποστηρίζουμε παρά τα προβλήματα που έχει ε, ε, ε, φέρνει για πρώτη φορά στην Ευρώπη μετά από πολλές αντιστάσεις κοινά όρια για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακου για τα βαριά επαγγελματικά οχήματα που συμβάλλουν κατά 6% στις συνολικές εκπομπές της Ένωσης, εκπομπές που προβλέπεται να αυξηθούν. Πέρα των target στόχων που είναι φιλόδοξοι αλλά μπορούμε να, τα, να τους πετύχουμε, έχουμε μια σειρά πρότυπων επιδόσεων στο δρόμο με εκπομπές για την κατανάλωση σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Αυτά τα πραγματικά στοιχεία συχνά απομακρύνονται από αυτά που περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά των εργαστηρίων και είναι αναγκαία για να αποφύγουμε στρεβλή συμπεριφορά και τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τρίτους για ελέγχους, για ανεξάρτητους ελέγχους. Κατά σημαντικό είναι το αίτημα της Επιτροπής μιας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της, της, ε, ε, των εκπομπών των οχημάτων αυτών σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωή τους. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης ένα μηχανισμό κινήτρων για την διάδοση ηλεκτρονικών φορτηγών ή χαμηλής, χαμηλών εκπομπών για να εξασφαλίσουμε από το 2025 ένα υποχρεωτικό ελάχιστο ποσοστό των οχημάτων αυτών ε, στο ύψος του 2%. Θα δοθούν κίνητρα σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και υποδομές για, την ηλεκτρική, για τα ηλεκτρικά φορτηγά. Στην πορεία για την ε, απομάκρυνση από τον άνθρακα, που κατά 94% εξαρτάται ακόμα και τώρα από το πετρόλαιο, θα πρέπει να εξετάσουμε και το ρόλο του φυσικού αερίου. Είναι αναγκαίο ωστόσο η Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ταμείο για την ε, ε, επανακατάτηση των εργαζομένων στον κλάδο για να καταστήσουν την βιώσιμη, τη μετάβαση βιώσιμη και κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Ο κόνισμος αυτός αποτελεί ένα επιπλέον βήμα σε μια Ευρώπη που αλλάζει προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στη συμμαχία μεταξύ βιομηχανίας και περιβάλλοντος. Ο κ. για λεπτό. Αύριο το μεσημέρι έχουμε την τελευταία ε, ψηφοφορία της τρέχουσας θητείας και πάλι έχουμε την ευκαιρία να ψηφίσουμε για συγκεκριμένα μέτρα στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για τα φορτηγά είναι ευθύνονται για 6% των συνολικών εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ένα τέταρτο συγγνώμη, των ε, οδικών μεταφορών. Και αυτές οι εκπομπές αυξάνονται ακόμα και στη δική μου χώρα, στη Φλάνδρα. Θέλουμε, αν θέλουμε λοιπόν ε, να πετύχουμε τους στόχους μας και τις δεσμεύσει μα για το κλίμα, θα πρέπει να πρασινίσουμε τον στόλο μας. Έχουμε την τεχνολογία αυτή. Είναι κρίσιμη σημασία, καταρχά ε, να υπάρξει ένα πρότυπο μείωση του διεξιδίου του άνθρακα για τα φορτηγά και τα κίνητρα για να ενθαρρυνθούν τα φορτηγά χαμηλών εκπομπών. Είναι σημαντικό και γι' αυτό λοιπόν το κόμμα μου το ΕΝΒΑ υποστηρίζει αυτή την τελική νομοθεσία, παρά το γεγονό ότι θα θέλαμε πιο υψηλό επίπεδο φιλοδοξία. Το πρασίνισμα λοιπόν του στόλου είναι πολύ σημαντικό για καλύτερη ποιότητα της ατμόσφαιρας, γιατί αυτή προκαλεί θανάτους πρόωρους. Τα πρότυπα αυτά φροντίζουν να υπάρχει και μείωση ε, του κόστου των καυσίμων. Αυτό είναι καλό για το καταναλωτή. Και τέλος, ε, η φιλόδοξη αυτή θέση προτύπων ε, χρειάζεται για να προσελκύσουμε επενδύσει και κοινοτομία, γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω από τι ΗΠΑ και την Κίνα. Ο για δύο λεπτά έχει το λόγο από την Άλτα. Πρόεδρε, ξεκινώ ευχαριστώντας τους συντρόφους και συναδέλφους που δούλεψαν μαζί μου αυτά τα χρόνια στις διαπραγματεύσεις. Είχα συνεργαστεί με τον κύριο Άικχαουτ και τον Κρίστο Φιέλνερ. Γκρίζαν τα μαλλιά του, είπε ο κύριος Φιέρνερ, αλλά αν δω τον επίτροπο ή και εμένα στον καθρέφτη θα έλεγα πολύ περισσότερα γκρίζα μαλλιά έχουν άλλοι. Έχουμε μπροστά μας κάποιες σημαντικές προκλήσεις. Πρώτον, κατακαιρματισμός στην κατασκευαστική διάσταση. Πολλοί κατασκευαστές θα τηρήσουν τους στόχους χωρίς δυσκολία, άλλοι θα το πετύχουν πολύ πιο δύσκολα και θα δυσκολέψουν έτσι τα πράγματα. Άλλο πρόβλημα είναι τα οχήματα μηδενικών εκπομπών, όπως τα λέμε. Τα αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών, αλλά με βρώμικο ηλεκτρισμό, δεν είναι και πολύ καθαρά. Πρέπει να έχουμε λοιπόν σημαντικούς στόχους, ε, όπως αυτούς που συζητήσαμε χτες με την Κρέτα Τούμπεργκ. Αν θέλουμε θα πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον σε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι ο δρόμος μπροστά. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε μια γέφυρα για το μέλλον με εναλλακτικά καύσιμα, εξασφαλίζοντας ότι οι εκπομπές, ε, τα όρια των εκπομπών είναι χαμηλότερα από αυτά του ηλεκτρισμού που χρησιμοποιούμε σήμερα. Η μεγαλύτερη πρόκληση προς τα εμπρός έχει να κάνει με αυτό που είπε στο ξεκίνημα της παρέμβασή του ο την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής τα επόμενα έτη. Μιλάμε τώρα για το επόμενο κοινοβούλιο, το οποίο θα έχει έτοιμη δουλειά, εξασφαλίζοντας ότι η πρόταση αυτή θα φτάσει στην, ε, τον προορισμό που έχει και ότι η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι θα γίνονται τα σωστά πράγματα. Ο Μπάς και άλλοι που μπορεί να είναι εδώ θα μπορέσουμε αν θέλουμε να βοηθήσουμε την υλοποίηση αυτής της, ε, ε αυτής της Κάποιο ε, ζητάνε να δέξει να απαντήσετε μια μπλε κάρτα. Πάντα με χαρά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον συναδελφό, τον κύριο Τορβάλτσε, γιατί το διοξείδιο του ανθρακά προφανώς και αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Και γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να δούμε και το κύκλο, σε όλο τον ε, κύκλο παραγωγής των φορτηγών και εδώ παίζει μεγάλο ρόλο και τι γίνεται με τα χρησιμοποιημένα φορτηγά. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα διαρκές ε, τέτοιο ζήτημα στις ε, πόλεις και αυτά θα μπορούσαν να έχουν μεγάλη συμβολή στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση αυτή. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό σημείο το οποίο χρειάζεται δεν είναι τόσο τα ευφύ οχήματα, αλλά κυρίω η ευφύ οδηγή. Δεν ξέρω πού μπορεί να βρει φυσικά ο κύριο Ρούμπι ευφύ οδηγού. Αλλά αυτό χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να μας ε, εκπαιδεύσουν στην οδήγηση. Χρειαζόμαστε τα τεχνικά εργαλεία για να έχουμε την κατάσταση υπό έλεγχο και να μην φοβόμαστε την τεχνολογία και όλες τις ευκαιρίες που παρέχει. Αν δεν φοβόμαστε, θεωρώ ότι μπορούμε να σώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, ο κύριος Εκ. 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Συχνά άσκησα κριτική στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά ε, τις αποφάσεις προς όφελος των μεγάλων ομίλων και προς ε, εις βάρος ε, της, του ανθρώπου, των, ζώων και του περιβάλλοντος. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος με αυτά που πέτυχε ο εισηγητής, ο κύριος Αικχάουτ. Αύριο θα ψηφίσουμε για τον πρώτο κανονισμό για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από τα φορτηγά. Παρά τις μεγάλες αντίδρασεις της, του οικονομικού κλάδου και πολλών κυβερνήσεων και κυρίω τη γερμανική κυβέρνηση, αυτή η πρόταση ξεπερνά κατά πολύ την αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντο. Δεν επαρκεί, ασφαλώ. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά να κάνουμε σε πολλού τομεί. Σήμερα είναι η τελευταία μου ομιλία αυτή εδώ στην Ολομέλεια. Δεν πρόκειται να είμαι βουλευτή στην επόμενη θετία. Θα σας καλέσω λοιπόν να τηρήσουμε το άρθρο 13 της Συνθήκης Λισαβόνας και να λάβουμε υπόψη την ευημερία των ε, δισεκατομμυρίων ζώων τα οποία τη χάνουν εκμετάλλευση και ε, τα θανατώνουμε, να κάνετε πολιτική με την καρδιά σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κλείσετε φυσικά και το κουμπί της λογικής. Θα πρέπει να αλλάξουν τα πολιτικά παράδειγματα. Να μην κοιτάμε μόνο την οικονομική ανάπτυξη, να μην είναι μόνο αυτό ο απότερο στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η ευημερία, η ευτυχία όλων των ε, ζώων, των οργανισμών και των ζώων. Αυτό αναμένουν οι πολίτε από εσά. Αυτό προσδοκούν οι πολίτε από εσά. Σα ευχαριστώ. Να είστε καλά και να έχετε το χέρι στην καρδιά στι μελλοντικέ πολιτικέ αποφάσει. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε Υπάρχει μια μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Ο κύριος Λίζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αξιότιμη κυρία συναδελφέ, κυρία Εξ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερα για το μέλλον προσωπικά. Έχω μία ερώτηση όμως να σας κάνω παρόλα αυτά. Αυτές τις πληροφορίες, από πού τις έχετε πάρει ότι αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας ξεπερνούν κατά πολύ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό ζήτησε και η γερμανική κυβέρνηση 15% και 30%. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ εύστοχος ο στόχο και δεν ξεπερνά την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Σέκα. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξή ότι σε κάποια σημεία στις διαπραγματεύσει πετύχαμε στόχους οι οποίοι ξεπερνούν ε, σίγουρα κατά πολύ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό το οφείλουμε κυρίως στον πολύ καλό συνάδελφό μα, τον εξαιρετικό συνάδελφό μα, τον κύριο Έκα, ο οποίο ε, πολέμησε με νύχια και με δόντια προκειμένου να είναι φιλόδοξη η έκθεση. Και γι' αυτό θα ήθελα προσωπικά να του απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για τους πράσινους, Ντέλη. Η κυρία Ντέλη έχει το λόγο. Παρακαλώ, Καρίμα. Συνάδελφοι, αυτή την εβδομάδα δεχθήκαμε στο Κοινοβουλίο την Κρέτα Τούμπεργκ που ήρθε να μας πει αναλάβετε δράση, κάντε κάτι, κάντε κάτι τώρα. Φροντίστε ότι εσείς που αποφασίζετε να επιτρέψετε να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να ζήσουν ευτυχισμένες σε έναν φιλόξενο κόσμο. Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τον πλανήτη και την υγεία μας, θα πρέπει να, και να μειώσουμε την ρήπανση, θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη και να υποχρεώσουμε τον κλάδο των μεταφορών να συμβάλλει όπως οι άλλοι. Στους δρόμους της Ευρώπης 5% ε, είναι μόνο τα φορτηγά μεταξύ των οχημάτων που παράγουν ωστόσο το 27% το 1 τέταρτο δηλαδή των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα των οδικών μεταφορών στην Ένωση. Αν θέλουμε μια μέρα να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις του COP21 να σώσουμε, για να σώσουμε το κλίμα και τον πλανήτη είναι καιρός να σταματήσουμε με αυτή την ανισορροπία. Με το κείμενο που υποβάλλεται ψηφίζουμε και κάνουμε τα πρώτα βήματα για την μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, λιγότερα ε, ε, αέρια μέχρι το 2000, με μείον 15% για τα φορτηγά. Ο κανονισμός πάει παραπέρα από την πρόταση επιτροπή και για πρώτη φορά δεσμεύει την Ευρώπη να μειώσει την ε, ρήπανση των μεγάλων φορτηγών. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι νικήσαμε. Τι δείχνει αυτή η νίκη. Δείχνει ότι όταν εμείς οι ψηφοφόροι Ακούμε τα αιτήματα, ιδίως της νεολαίας, που κάθε εβδομάδα κάνει απεργία για να σώσει το κλίμα. Όταν εγκρίνουμε ε, όταν περνάμε από τα ωραία λόγια σε συγκεκριμένες δράσεις μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Προσοχή ωστόσο. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε την δυνατότητα τα παιδιά μας να ανασάνουν, να ζήσουν ελεύθερα, να χαρούν αυτό τον ωραίο πλανήτη, θα πρέπει αύριο να ψηφίσουμε το κείμενο αυτό, γιατί ψηφίζοντας το κείμενο ψηφίζουμε για το κλίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ για την Ευρώπη των Εθνών και Ελευθεριών. Λαντσίνη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κλάδος της κίνησης είναι θεμελιώδης και για την οικονομία και για την κοινωνία των κρατών μελών. Ωστόσο εδώ συνεχώς ξεχνάμε αυτή τη διάσταση και δεν ακούμε τα αιτήματα των επιχειρηματιών και εργαζομένων. Τα μέτρα που περιλαμβάνει η πρόταση αυτή είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων αναχρονιστικά ή, ε, παράλογα. Μιλάμε για μια βιώσιμη μετακίνηση προς την κινητικότητα χωρίς κατανάλωση, χωρίς όμως να κάνει μια αξιολόγηση των αντικτύπων των μέτρων που προτείνονται. Το μέτρο μιλά, υποχρεώνει να στραφούμε στα ηλεκτρικά, εξαφανίζοντας και αγνώντας τις άλλες εναλλακτικέ λύσεις που υπάρχουν στην αγορά. Θα έπρεπε εξ αρχής να προβλέπεται η χρήση μείγματος τεχνολογιών και μεγαλύτερες προθεσμίες για να διευκολυθούν οι επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών εκπομπών ε, μπορεί να βελτιωθεί σε σχέση με τα υπόλοιπα οχήματα, ιδίως ό,τι αφορά τα ε, μεγάλα τα Ο κλάδος θα πληγεί εις βάρος της ευρωπαϊκής ε, και των κρατών μελών. Η Ευρώπη θα γίνεται ακόμα περισσότερο ε, εξαρτημένη από τρίτες χώρες για την απακτήση ε, μπαταριών. Και Επιπλέον, όπως αναφέρει ο τύπος και παράδοξα, χρησιμοποιήθηκαν μόνο ε, νέες στήλε για ε, ηλεκτρική ενέργεια που όμως τροφοδοτούνται από δίζελ. Ε, ο κλάδος της, της, της οδικής κίνησης θα μπορούσε να χάσει ε, μόνο στη Γερμανία μεταξύ 75.000 και 210.000 ε, μονάδων μέσα στο 2030. Σκεφτούμε καλύτερα την πρόταση αυτή που όπως διατυπώνεται αυτή τη στιγμή στην ουσία είναι ακατανόητη και με αποτελέσματα αντίθετα από αυτά που έχει θέσει ως στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σόσνιετς. Ένα λεπτό. Ε, στα έγγραφα μιλάμε συνεχώς για μηδενικές εκπομπές, αλλά μηδενικές εκπομπές δεν υπάρχουν ούτε θα υπάρξουν. Είναι ένα εργαλείο marketing που χρησιμοποιείτε εσείς ή αυτοκινητοβιομηχανίες. Μεταφορές μηδενικών εκπομπών δεν είναι δυνατές. Κάποιο σε, ε, Κάποιο θα εκπέμπει. Αν δεν εκπέμπουν τα οχήματα, θα εκπέμπουν οι βιομηχανίε οι οποίε θα παράγουν την ενέργεια που χρησιμοποιούν τα οχήματα. Οπότε πολύ ωραία να δράσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή η τεχνολογία δεν μας επιτρέπει να φτάσουμε σε μηδενικές εκπομπές. Κάπου θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια και θα χρειαστεί να μεταφερθεί. Μηδενικές εκπομπές δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν η έκθεση αυτή είναι ανεύθυνη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Λίζα. Ενάμιση λεπτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Και είναι πολύ καλό το γεγονό ότι αύριο για πρώτη φορά ορίζουμε όρια για τι εκπομπέ των βαρέων οχημάτων. Γιατί όλοι τα μίστα πρέπει να συμβάλλουν αυτό που του αναλογεί στη μείωση των εκπομπών. Είναι φιλόδοξο αλλά εφικτό το σχέδιο που έχουμε μπροστά μα. και είναι καλό που έχουμε που δεν υποκύψαμε στις υπερβολικές ε, ε, απαιτήσει των πράσινων στο κείμενο αυτό. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μπαθ για την ε, ρεαλισμό που έδωσε, γιατί ήθελε πολλά παραπάνω αρχικά, αλλά επικεντρώθηκε στα ουσιαστικά και αυτό ήθελε και το ΕΛΚ, αυτό ήθελε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν ευφυέ αυτό. Να ευχαριστώ και τον Κρίσταφερ Φιέρνερ για την δέσμευσή του, όχι μόνο για το θέμα αυτό, αλλά και για πολλά άλλα θέματα. Αλλά θα ήθελα να πράξω την ευκαιρία όλος ιδιαίτερος για να ευχαριστήσω και τον Επιτρόπο κύριο Κανιέτα, γιατί στην ακρόαση, ακρόαση του αντιμετώπισε τα πειρά της κριτικής και τότε ακόμα και αυτοί που τον επέκριναν τότε θα πρέπει σήμερα να ομολογήσουν ότι πετύχαμε πολλά μαζί για την προστασία του κλίματος στην Ευρώπη και είναι η τελευταία νομοθεσία που θα περάσει το Κοινοβούλιο αυτό. Γι' αυτό να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον Επιτροπό, τον κύριο Κανιέτε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε και ένα θέμα νομίζω που θα χαρακτηρίσει την επόμενη περίοδο είναι η ενίσχυση των συντροδρόμων. Καλό είναι να ρυθμίσουμε και τα φορτηγά, αλλά θα πρέπει όλο και πιο πολλά εμπορεύματα και ε, επιβάτες να μεταφερθούν στο συντροδρόμο και να δούμε ότι σε ό,τι αφορά την ε, μείωση των εκπομπών είναι πολύ πιο επιβαρημένος ο συντροδρόμος από ότι οι άλλοι τομείς μεταφορών. Και εδώ θα πρέπει κάτι να κάνουμε λοιπόν στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και κύριε Λίζα, έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Σόσνη, έτσι. Την αποδέχεστε βεβαίω. Με χαρά. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρο. Πολλά πατήχαμε. Πετύχαμε σε ό,τι αφορά το κλίμα σε ό,τι αφορά κάποια στερεότυπα τα οποία πέρασαν στο κλίμα. Τι θα σημαίνουν όμως όλα αυτά συγκεκριμένα για το κλίμα, ο κύριος Λίζε. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά όταν ε, μου κάνετε την ερώτηση αυτή να σας το πω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πετύχει τους στόχους της για το 2030 και αποφασίσαμε λοιπόν για μια νομοθεσία και αύριο θα αποφασίσουμε το τελευταίο τμήμα της νομοθεσίας αυτής, όπου ο νομοθετικός πώς δημιουργούμε τους όρους για να εκπληρώσουμε και με το παραπάνω τους στόχους μας για το 2040. Είναι απαραίτητο λοιπόν η Ευρώπη να αποτελέσει πρότυπο και για τις άλλες επίρρους και παράλληλα έχουμε και κανόνες που δεν θα διώξουν τη βιομηχανία από την Ευρώπη. Θεωρώ ότι αυτό είναι καλή ισορροπία και όταν έχουμε τα βέλη τη κριτική και από τι δύο πλευρέ του πολιτικού φάσματο, αυτό είναι καλό δείγμα ότι είναι ισορροπημένη η νομοθεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ντάλη για 1,5 λεπτό. Μυρία, μου, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και θα ήθελα καταρχά να συγχαρώ τον εισηγητή μα, τον κύριο Άικχαουτ, για τη δουλειά που έκανε και το συμβιβασμό που πέτυχε, γιατί ξέρω δεν ήταν εύκολο ο φάκελο αυτό. Ήταν πάρα πολύ θετικό το γεγονό ότι έχουμε πλέον άλλη μία πολιτική για τη μείωση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα όπου δεν είχαμε πρότυπα για τα ε, βαρέα οχήματα. Παρά το γεγονό ότι γνωρίζαμε την μεγάλη επίπτωση που έχουν τα φορτηγά αυτά στην ε, παγκόσμια αύξηση του τη θερμοκρασία. Και αυτή αναμένεται να αυξηθεί. Έχει έρθει λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου να εγκρίνει δεσμευτικά πρότυπα η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση των εκπομπών. Ήταν λοιπόν δύσκολο το έργο αυτό. Η διαπραγμάτευση για το Συμβούλιο, με το Συμβούλιο για την θέση των benchmarks ήταν πραγματικά μεγάλο επιτεύγμα. Το ξέρω αυτό από προσωπική εμπειρία να ευχαριστήσω και τον εισηγητή από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, τον κύριο Τσόφολη, για την μεγάλη του δέσμευση και τον ρόλο που έπαιξε για να πετύχουμε συμβιβασμό. Η θέση του Κοινοβουλίου θέτει το σωστό επίπεδο φιλοδοξίας. Αυτό χρειάζεται για να ε, καταφέρουμε να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας για το κλίμα και πιστεύω ότι το μέλλον των καθαρών οχημάτων και των φορτηγών θα καθοριστεί από την κρατομία μόνο με ισχυρά κίνητρα για την παραγωγή οχημάτων χαμηλών εκπομπών και μηδενικών εκπομπών τελικά θα περάσει την αλλαγή αυτή. Αυτό αποτελεί το σκόπο μας και το στόχο μας. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε με τη δουλειά μας και προσβλέπω και τις μελλοντικές μας προσπάθειες τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο λόγος στην συνάδελφο εγώ Νταλόντα για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε. Επιτέλους ε, καθορίζονται ε, στόχοι μείωση ε, εκπομπών για τα, βόρεια, για τα βαριά οχήματα. Τέτοιου είδου ε, στόχου και πολύ πιο φιλόδοξου είχαμε στηρίξει εμεί στην Επιτροπή Μεταφορών. Όμω η Γερμανία και άλλε χώρε, πιεσμένε από την αυτοκινητοβιομηχανία του, μείωσαν του ε, στόχου. Παρ' όλα αυτά, οι εκπομπέ διοξείδου του άνθρακα συνεχώ αυξάνονται τα τελευταία χρόνια στι οδικέ μεταφορέ. Αντίθετο, η αναθεώρηση του 2022 θα είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να προσαρμόσουμε την νομοθεσία και ενδεχομένως να καλύψουμε περισσότερους τύπους οχημάτων και ενδεχομένως να ξαναδούμε τους στόχους μας. Παρόλο ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλης από τα κράτη-μέλη, χαίρομαι που αυτή τη στιγμή έχουμε ένα οδικό χάρτη υποχρεωτικό. Ο κανονισμός αυτός είναι ένα βήμα για να καταπολεμήσουμε την ατμοσφαιρική μόλυνση και να σεβαστούμε τους κλιματικούς στόχους, ιδιαίτερα του Παρισιού, που θα περιορίσουν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Αυτό προς όφελος των επόμενων γενιών. Η Ευρώπη δρά με συγκεκριμένο τρόπο κατά της μόλυνσης. Και τελευταία μου αυτή ομιλία στην Ολομέλεια θέλω, να υπογραμμίσει ακριβώς αυτή την πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Catch the eye. Δύο αιτήματα έχουν ε, γίνεται, έχουν υποβληθεί. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Εκχάουτ και όλους τους συναδέλφους ε, που βοήθησαν να θέσουμε τέτοιους φιλόδοξους στόχους για τα βαρέα οχήματα. Επίσης να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας για διαφορετικά χαρτοφυλάκια, διαφορετικούς φακέλους ε, που έχουν σχέση με τους στόχους του Παρισιού, την κυρία Ντάλη πιο συγκεκριμένα ε, είχαμε κάνει πρόταση για πιο φιλόδοξους στόχους και ελπίζουμε ότι αυτές οι προτάσεις, ε, οι προτάσεις του ΕΛΚ ε, βοήθησαν. Προφανώς η κλιματική αλλαγή υπάρχει. Πρέπει να προστατεύσουμε τα οικοσυστήματά μας και να μειώσουμε την τοξικότητα της ανθρώπινης δράσης στον πίνακα. Οι επιστήμονες στέλνουν σήμα κινδύνου στην κοινωνία. Αλλά ε, υπάρχει κάτι το οποίο κάνουμε, ε, δεν κάνουμε σωστά. Δεν προχωράει αρκετά γρήγορα η μείωση της χρήσης του ε, άνθρακα. Κέλλη, Σον, e έχεις το λόγο. ασχολούμαι με θέματα κλιματικά καθ' όλη τη διάρκεια της αιτίας. Και χαίρομαι για την πρόοδο που κάναμε στο Κοινοβούλιο. Συγχαρητήρια στον Επίτροπο Και τον κύριο Έκχαουτ, που αποτέλεσε ατμομηχανή σε αυτό το τομέα τα τελευταία πέντε χρόνια. Όπως είπε η Μύρια Μτάλη, ε, έχουμε πλέον μια πολιτική για τα βαρέα οχήματα. Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές. Όσο βελτιώνεται η οικονομία, ε, εγώ πηγαίνω από το, το, σπίτι μου στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου και από το Στρασβούργο στη Φραγκφούρτη και βλέπω όλο και περισσότερα βαρύ οχήματα στους δρόμους. Η μείωση αυτή που προβλέπουμε δεν σημαίνει ότι θα, μειώσει, θα μειωθούν οι μεταφορές. Απλά θα τις κάνει πιο ενεργειακά αποδοτικές. Οπότε μπορούμε να γίνουμε πιο φιλόδοξοι τα επόμενα χρόνια, αλλά είναι μια καλή αρχή. Είναι μια λογική πρόοδος, προοδευτική, σταδιακή και νομίζω με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουν το περιβάλλον μας. Συγχαρητήρια σε όλους. Thank you διαδικασία του Κατσδιάη. Το λόγο τώρα για την Επιτροπή ο Επίτροπος Άρια Κανιέται. Παρακαλώ κύριε Επιτροπέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι βουλευτές για τη συζήτηση αυτή. Να απαντήσω σε μια απευθείας ερώτηση που μου έφεσε ο κ. Σόσνιεκ. Ρώτησε, τι έκανε αυτό το κοινοβούλιο για την αργή του κλίματος. Η απάντηση μου είναι πολλά. Τι έκανε, είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλλαγή του κλίματος. Όχι πολλά. Πριν το 2020 θέσαμε στόχους μείωσης των εκπομπών και το 2017 μειώσαμε τις εκπομπές κατά 17% σε σχέση με το 1990. Μειώσαμε τις εκπομπές, αναπτύξαμε, αναπτύξαμε τα ανανεώσιμα, κάναμε καλύτερη ε, λειτουργία των επιδόσεων, αλλά το κοινοβούλιο αυτό διπλασίασε το πλαίσιο για την ενέργεια. Ήμουν στην πολιτική, είμαι στην πολιτική 38 χρόνια, έχω έχω, έχω υπηρετήσει σε εθνικά, περιφερειακά και ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Ποτέ δεν είδα τόσο έντονη νομοθετική διαδικασία ε, δραστηριότητα όσο εδώ. Και θέλω να ευχαριστήσω τους προέδρους των Επιτροπών, την κυρία Βάλη, τον κύριο Μπούσεκ, τον Τζοβάνι Λαβία, όλους τους εισηγητές, ξεκινώντας από τον κύριο Άικχαουτ, που έκανε εξαιρετική δουλειά που ήταν και δύσκολο σε κάποιες περιπτώσεις όπως στα ανανεώσιμα. Και αυτό που κάναμε είναι ότι υιοθετήσαμε πολλά νομοθετικά κείμενα που θα οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών το 2030 κατά 45% και αν αλλάξουν και θα αλλάξουν το 2030 θα έχουν 60% μειώσεις των εκπομπών, με μεγάλο πακέτο. Και ένα από τα πιο σημαντικά είναι ο μέσος, το μέσο ποσοστό πολιτικών, πολιτικής υποστήριξης προτάσεις αυτές. Στο πακέτο ενέργειας 80% των ψηφοφοριών ήταν υπέρ. Στο κλίμα 76%. Σημαντική λοιπόν πολιτική υποστήριξη για την νομοθεσία που υιοθετήσαμε το 2030 που σημαίνει ότι Είχαμε έναν διάλογο, υπήρχε αμοιβαία κατανόηση, υπήρχαν διαπραγματεύσεις και όπως σας είπα ήταν μια απίθανη ευκαιρία. Μετήσχα σε 71 τριμερείς διαλόγους. Δύσκολους που πάνω από 350 ώρες της ζωής μου. Αλλά ήταν εξαιρετικές ευκαιρίες για να μάθω και να σας ευχαριστήσω όλους γιατί η δουλειά αυτή ήταν μια εξαιρετική δουλειά που δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την δική σας εμπλοκή. Εσείς πιέζετε και εμείς ε, απαντάμε. Αυτό είναι ο θεσμικός ρόλος του καθενός. Το βασικό στοιχείο είναι ότι περνάμε ένα κείμενο που θα εφαρμοστεί για την επόμενη 20 ετία, αλλά έχουμε τη δυνατότητα αναθεώρησης καθοδών για με αύξηση των στόχων. Στις 77% των πιθανών ψηφοφόρων για τις ευρωεκλογέ ανέφεραν σε μια σφιγμομέτρηση την περασμένη εβδομάδα ότι το περιβάλλον ήταν ο βασικός λόγος να πάνε να ψηφίσουν τι ευρωεκλογέ. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Η αλλαγή του κλίματος είναι ένας βασικός παράγοντας για να συζητηθεί στις Ευρωεκλογικές. Σας παροτρύνω να κάνετε δύο πράγματα. Πρώτον, να εξηγήσετε στους πολίτες της Ευρώπης τι κάναμε αυτά τα πέντε χρόνια. Και επίσης, να πείτε τι θέλετε να κάνετε τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό θα φέρει περισσότερο κόσμο στις κάλπες και θα μπορέσει το Κοινοβούλιο στην επόμενη θητεία να βοηθήσει την ολοκλήρωση του πακέτου, την περαιτέρω πρόοδο και την συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων για να μπορέσει η Ένωση να γίνει το 2020 η πρώτη μεγάλη οικονομία που θα είναι ε, ε ενεργειακά ουδέτερη. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα ο κ. Σάικα, ο εισηγητής. Μπάς, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και καταρχά, μια και βρισκόμαστε σε τέτοια κλίμα ευγνωμοσύνη, να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο, τον Επίτροπο Μαρία Κανιέτα, για τη δουλειά που έκανε. Και προφανώ και είχαμε στιγμέ όπου διαφωνήσαμε και κάποιε από τι ώρε αυτέ τι ε, περάσαμε μαζί. Να πω ότι Ανά πάσα στιγμή ο διάλογο ήταν καλό. Δεν συμφωνούσαμε πάντα, αλλά υπήρχε πάντα αμοιβαίο σεβασμό και αυτό είναι απαραίτητο για το μέλλον. Και έχετε απόλυτο δίκιο ότι πετύχαμε πολλά. Πετύχαμε πολλά για το κλίμα, για την ενέργεια, για την κινητικότητα. Δεν έχουμε ολοκληρώσει όμω το έργο μα. Και αυτό, όπω είπατε, δεν έχουμε ακόμα ε, μπει στη σωστή τροχιά για την ε, ε, οικονομία τυφλική προ το κλίμα. Και αυτό θα το τονίσουμε και αύριο. Και είναι ένα από του λόγου αυτού για του οποίου αύριο και στις ευρωεκλογέ. Το θέμα θα είναι το κλίμα, θα είναι οι εκλογές του κλίματος. Και να σας πω, δυστυχώς να δώσω και ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ξαναήλθατε, γιατί μπορώ να σας απαντήσω για το που εμείς ως Κοινοβούλιο κάναμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιο φιλόδοξη. Καταρχάς, ο, ο στόχος για το 2030 πλέον είναι νομικά δεσμευτικός. Αυτό δεν ήταν στην αρχική πρόταση. Πολύ σημαντικό, γιατί είναι σαφές μήνυμα για το που οδεύουμε. Δεύτερον, κλείσαμε πολλά παραθυράκια στις προτάσεις και κυρίως αυτά για τις ε, τα υπερπιστωτικά μόρια σε ό,τι αφορά τα ε, οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και τρίτων ε, σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα για τα οχήματα στον δρόμο, τα βελτιώσαμε για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε ότι αυτά που συμφωνούμε θεωρητικά θα εφαρμοστούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά τον Dieselgate. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι τόσο απαραίτητα και τόσο κρίσιμα πέρα από τι τεχνικέ βελτιώσει και τι ρήτρε αναθεώρηση και το καθεξή. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι τόσο σημαντικά λοιπόν που στέλνουν ένα μήνυμα προ του επενδυτέ, του κατασκευαστέ ότι το μέλλον θα είναι μηδενικέ χαμηλέ εκπομπέ στα οχήματα και ότι αν συνεχίσουν όπως ε, σήμερα δεν θα πάνε μπροστά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναγκαστικά λοιπόν καταλαβαίνετε. Σα έδωσα τις απαντήσει αυτέ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ. Προσβλέπω στην αυριανή ψηφοφορία να δούμε τι θα μπορέσουμε να πετύχουμε και μετά. Εν ώψη και τη Συνόδου στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο, γιατί περιμένω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει τι ε, εθνικέ τη ε, σύνδρομες βλέπω να προσεύχεται και ο Επίτροπος να ευχηθώ και εγώ για αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Πέρα στη συνδρίαση. Και θα γίνει αύριο η ψηφοφορία. Βάσει τη ημερήσια διάδοξη προχωρούμε τώρα στην ε, έκθεση Γκαζίμπ για την πρόθεση καθαρών και ενεργειακών αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών. Δίνω αμέσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Γκαζίμπ για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε, κύριε Επίτροπε. Πρόκειται για μια οδηγία που θα στηρίξει τα οχήματα, ε, τα ενεργειακώς πιο αποδοτικά οχήματα. Το 60% Ορισμένοι λένε 65-66% της μόλυνσης ε, στις πόλεις λέγεται ότι οφείλεται στον τομέα των μεταφορών. Μπορούμε να βελτιώσουμε τα οχήματά μας, ε, τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, τα φορτηγά, αλλά υπάρχουν εκπομπές και από αλλού. Και αυτό το βλέπουμε στους, στις κρατικές προμήθειες και στους δημόσιους διαγωνισμούς. Αν εγκρίνουμε αυτό το κείμενο, θα εγκρίνουμε πολύ φιλόδοξους στόχου. Και πρέπει αυτοί οι στόχοι να είναι εφαρμόσιμοι στην πράξη. Από τις δημόσιες διοικήσεις. Οπότε είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να στηριχθούν από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Οι στόχοι αυτοί λαμβάνουν υπόψη και τις δυνατότητες των διαφορετικών κρατών μελών. Ελπίζουμε να μπορούν να υλοποιηθούν και τα κράτη-μέλη να φτάσουν μέχρι σε αυτό το σημείο. Προφανώς δεν μιλάμε για το 100% των αγορών γιατί υπάρχουν παραδοσιακές τεχνολογίες, σημαντικές τεχνολογίες που δεν μπορούν να εγκαταλειφθούν από τη μια μέρα στην άλλη. Οι τοπικές αρχές μας είπαν ε, για παράδειγμα ότι τα υβριδικά οχήματα είναι μια καλή βοήθεια για να μειωθούν οι εκπομπές και να προχωρήσουμε προς μηδενικές εκπομπές. Υπάρχει μια τεχνογνωσία που ήδη είναι γνωστή για αυτά τα οχήματα. Χρειάζεται επίσης να εξασφαλίσουμε μια ελαστικότητα μέσω της ε, οδηγίας για τα εναλλακτικά καύσιμα, για παράδειγμα, πρόκειται για κείμενα τα οποία ήδη υπάρχουν. Το κείμενο αυτό αφορά και τα βαρέα και τα ελαφρά οχήματα και θα επηρεάσει και τα λεωφορεία στις δημόσιες μεταφορές. Οι περισσότερες αγορές γίνονται μέσω κρατικών διαγωνισμών, οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η οδηγία. Η, τα αυτοκίνητα είναι ο βασικός στόχος αυτής της οδηγίας, μπορώ να πω και οι κατασκευαστές των λεωφορείων έχουν πλέον τεχνολογία την οποία θα πρέπει να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο και να την χρησιμοποιήσουν προκειμένου τα νέα λεωφορεία να μπορούν να ανταγωνιστούν στις παγκόσμιες αγορές, όχι μόνο στην ευρωπαϊκή αγορά. Για παράδειγμα, η, ε, εταιρεία Solaris στην Πολωνία έχει λεωφορεία με μηδενικές εκπομπές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης. Ελπίζουμε ότι η τεχνολογία ε, χαμηλών εκπομπών η οποία αναπτύσσεται με τη χρήση βιομεθανίου για παράδειγμα θα επιτρέψει να μειωθούν οι εκπομπές ε, στις ε, δημόσιες μεταφορές. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εποχωρηθούμε καλύτερα από το βιοαέριο, τα βιοκάψιμα Κάτι το οποίο θα είναι πολύ θετικό για το περιβάλλον μας. Το βλέπετε αυτό στην πρότασή μου. Στο μέλλον θα κατασκευάζονται οχήματα μηδενικών εκπομπών. Αυτό το ξέρουμε. Και οι τεχνολογίες βελτιώνονται. Όμως θα πρέπει να δούμε τις τεχνολογίες αυτές στο σύνολό τους. Για παράδειγμα, μπαταρίες και συσσωρευτές. Και αυτοί επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον, το βλάπτουν. Οπότε θα πρέπει να γίνει η, μείωση να γίνει ε, οριζοντίως. Ε, πρέπει να μειωθεί η μόλυνση του περιβάλλοντος και από τις μπαταρίες, να μπορούν να ανακυκλωθούν κλπ. Επίσης, να μπορούν να χρησιμοποιούν οι μπαταρίες λιγότερους ε, μολυσματικούς παράγοντες. Θα πρέπει να δώσουμε με αυτόν τον τρόπο μια όθηση στις ε, ευρωπαϊκές εταιρείες για βελτιωμένες απόδοσης μπαταρίες και πιο καθαρές μπαταρίες. Η αυτοκινητοβιομηχανία με την κατάλληλη έρευνα και καινοτομία θα παράγει αυτοκίνητα, οχήματα τα οποία πραγματικά θα είναι πολύ πιο αποδοτικά και πολύ πιο χρήσιμα. Ε, ευχαριστώ πολύ όλους και όλες τους συνεισηγητές και όλους Είχαμε μερικά προβληματάκια, αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό. Ευχαριστώ πολύ και την Κομισιόν που στις δύσκολες στιγμές μας βοήθησε να βρούμε συμβιβασμούς. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Ρουμανική Προεδρία που μας βοήθησε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Για την Επιτροπή, η Επίτροπος. Πούλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καλωσορίζουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα με τη, μαζί σας την έκθεση Γκοζίμπ. Σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική δουλειά που έχετε κάνει. Και εσείς και οι συνηγικέ και οι όχι μόνο τώρα, αλλά σε όλη τη διαδικασία. Όπως είπατε, η συνεργασία δεν ήταν πάντα εύκολα, ήταν ανοιχτή, με αφοσίωση και με αποτελέσματα. Χάρη στην δέσμευση και την αποφασιστικότητα όλων των τριών εμπλεκόμενων στην νομοθεσία οργάνων είχαμε σωστό, καλό αποτέλεσμα. Ένα καθαρό πακέτο κινητικότητας. Ο, ο δημόσιος τομέας έχει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της απομάκρυνσης από τον άνθρακα στις μεταφορές. Η τα λεωφορεία κυρίως όπου οι δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν το 70% της αγοράς χρησιμοποιώντας ε, την, ε, τις δημόσιες συμβάσεις για την επιτάχυνση των καθαρών οχημάτων, η οδηγία επιτρέπει να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για, την μηδενι... για τη κινητικότητα μηδενικών εκπομπών. Κατά την άποψή μα, το κείμενο που συζητήθηκε στον τριμερή διάλογο στις 11 Φεβρουαρίου αντιπροσωπεύει μια καλή συμβαστική λύση μεταξύ των διαφόρων θέσεων και ε, ετοιμάτων. Δείχνει ότι υπάρχει επαρκή φιλοδοξία, αφήνοντα ε, αρκετή ευελιξία για την υλοποίηση, ούτως ώστε οι στόχοι της οδηγίας να μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς μεγάλο διοικητικό βάρος για τις δημόσιες αρχές. Με την, με την έγκριση της αναθεωρημένης οδηγίας δίνουμε ορισμό ότι είναι καθαρό όχημα και θέτουμε σαφείς στόχους για τις δημόσιες συμβάσεις, ιδίως ειδικού στόχους για λεωφορεία μηδενικών εκπομπών. Έχω εμπιστοσύνη στο ότι η συμφωνία που επιτεύχθη στον τριμερή διάλογο θέτει επαρκή, επαρκώς σαφή ορισμό και επαρκώς φιλόδοξους εθνικούς στόχους. Το κείμενο επίσης δίνει μεγάλη ευελιξία για το πώς οι προσπάθειες ε, επιμερίζονται μεταξύ κρατών μελών, επιτρέποντας μία κοστοποτελεσματική εφαρμογή που δεν θα δημιουργήσει σημαντική επιβάρυνση στις αρχές των κρατών μελών πολλές πόλεις μας, το Άμστερνταμ, το Βερολίνο, ε, η Βαρσοβία, το η Βαρκελόνη, το Μιλάνο, η Λουμπλιάνα, το Μόναχο και πολλές άλλες ήδη έχουν αναλάβει εθελούσες δεσμεύσεις ξεπερνώντας αυτό που απαιτεί η οδηγία. Θα βοηθήσουμε και άλλες πόλεις να ακολουθήσουν το παραδείγμα τους. Η αναθεώρηση θα επεκτείνει και το πεδίο εφαρμογή οδηγίε για να καλύπτονται δημόσιες ε, προμήθειε μέσω πρακτικών όπως ε, ε, ενοικίαση πώληση και σύντομη ενοικίαση. Αυτό θα αντικατοπτρίζει και τις καλύτερες πρακτικές των κρατικών προμηθειών, μειώνοντας τον αντίκτυπο στην αγορά. Από κοινού, τα μέτρα αυτά θα παράσχουν σαφή μηνύματα προς την αγορά επιτρέποντας τις αρχές, τους κατασκευαστές και τους επενδυτές να προγραμματίσουν καλύτερα την μετάβασή μας μέχρι τα μέσα του αιώνα στην κινητικότητα μηδενικής ε, εκπομπής, βελτιώνοντας την μείωση της συμμετοχής του άνθρακα στην κινητικότητά μας και την επίτευξη του μηδενικού στόχου το 2050. E Ευχαριστώ Επίτροπε. Για την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, Ντέλη. Έχει το λόγο που δεν είναι εδώ όμως. Αργότερα. Πολιτικές ομάδες. Ξεκινούμε από το ΕΛΚ. Ο κύριος Πίπερ έχει το λόγο. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση των επιζήμιων ουσιών ρυθμίζεται καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το σε εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την ε, αποδοτικότητα, την και τη μείωση των εκπομπών. Και έτσι λοιπόν εργαζόμαστε καλύτερα στον οικολογικό σχεδιασμό, στη συνεργική επισήμανση και σε πολλά άλλα θέματα συνεργαζόμαστε ευρωπαϊκά. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει τέτοια εγγύηση Είμαστε υπέρ των ευρωπαϊκών διατάξεων. Δεν θα πρέπει όμως να επισέλθουμε σε μεγάλο επίπεδο λεπτομερία και κυρίως όχι στους δήμους και στις κοινότητε να μπούμε να κάνουμε κομμάτι με τις διατάξεις αυτές ε, κυρίες και κύριε θεωρώ ότι ε, ανοίγουμε ένα μεγάλο πλήγμα στον κόλπο των ε, ε, δήμων και Κοινωνιτήτων, γιατί απέχουμε πολύ από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις για τα ηλεκτρικά ε, λεωφορεία. Κάνουν τις μεταφορές πολύ ακριβές και το πώς ε, ρυθμίζονται όλα αυτά. Θα πρέπει να τα αφήνουμε στο επίπεδο των τοπικό. Όχι να υπάρχουν ε, γενικές διατάξεις από τις Βρεξέλλες και στην πατρίδα μου θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση και δικαίως για την υπερβολική ανάμειξη των Βρυξελών και μεγάλο τμήμα του ΕΛΚ θα απορρίψει την οδηγία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Και το λόγο λοιπόν τώρα έχει από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες ο κύριος Ντάνς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Τη ευχαριστίας μου στον εισηγητή, τον κύριο Γκριπ, και την Κομισιόν. Το Συμβούλιο κρίμα δεν είναι εδώ. Εξαιρετική δουλειά που έχουμε κάνει. Κύριε Κρύπ, είσαστε πολύ δίκαιο ω συγητής, πολύ αμερόληπτος. Ε, διεξάγατε τις διαπραγματεύσει μεταξύ των διαφορετικών ομάδων με εξαιρετικό τρόπο. Συγχαρητήρια. Ο φάκελο αυτός είναι πολύ καλό παράδειγμα για το λόγο για τον οποίο έχουμε εκλεγεί εδώ και το ρόλο μας. Πρέπει να γίνουμε πιο δραστήριοι στον καθαρισμό των οχημάτων, στο να κάνουμε τα οχήματα που κυκλοφορούν στου δρόμου πιο καθαρά, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και γιατί ε, η ποιότητα γενικότερα του αέρα τη πόλη είναι πολύ κακή. Οι κρατικέ προμήθειε αντιπροσωπεύουν το 14% του ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το 45% των ε, λεωφορείων που κυκλοφορούν. Είναι λοιπόν πολύ σωστό και πολύ επίκαιρο που θα χρηματοδοτήσουμε τα πιο φτηνά, ε, πιο συγγνώμη, καθαρά οχήματα ε, μέσω των κρατών μελών. Το 2030 το 60% των λεωφορείων θα πρέπει να πληρούν τους όρους οδηγίας. Η Κομισιόν βέβαια και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι τοπικές αρχές θα έχουν τα κατάλληλα μέσα και επαρκείς πόρους. Απαντώντας στους συναδέλφους του ΕΛΚ, θα ήθελα να πω το εξής. Χρειαζόμαστε αυτή τη φιλοδοξία. Δεν μπορούμε να καθόμαστε στον καναπέ μα και να ελπίζουμε ότι τα πράγματα από μόνα του κάπω θα κινηθούν. Πρέπει να πάρουμε δύσκολε αποφάσει σήμερα. Σε όλα τα κράτη-μέλη βλέπουμε νέου να διαδηλώνουν, να διαμαρτύρονται και όχι μόνο νέου, γενικότερα ευαισθητοποιημένου πολίτε. Θα πρέπει να αντιδράσουμε τώρα. Και είμαι περήφανο που το κάνουμε. Το Κοινοβούλιο και οι πόλη είναι αυτέ που ζητούν πάντοτε περισσότερα, ενώ τα, οι κυβερνήσει, οι κεντρικέ κυβερνήσει είναι αυτέ που κρατάνε τα χαλινάρια. Αυτή είναι η εμπειρία μου τα τελευταία πέντε χρόνια. Ε, δεν ξέρω αν θα επιστρέψω στο κοινοβούλιο αυτό ω Βρετανό. Αν όμω αυτή είναι η τελευταία μου ομιλία, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είστε εδώ για να κάνετε το ορθό. Έμαθα πολλά από εσά και ελπίζω θα επιστρέψω για να μάθω περισσότερα. Thank you very much, dear colleague, and good luck. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Καλή τύχη σας εύχομαι. Και τώρα το λόγο έχει από το ECR ο κύριος Ντεμέσμακερ για 1,5 λεπτό. Μάρκα, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Επιτροπή, συνάδελφοι, πριν από λίγο συζητήσαμε για τι πρώτε μειώσει των διοξιδίτων ανθρακά για τα βαρέα οχήματα. Και τώρα έχουμε ένα φάκελο για τα καθαρά και ενεργειακώ αποβατικά οχήματα και πώ μπορούμε να τα προωθήσουμε. Είναι καλό το αποτέλεσμα και νομίζω πάρα πολύ σημαντικό ως μήνυμα για την τελευταία ε, ολομέλεια αύριο, την ψηφοφορία δηλαδή, τη τρέχουσα θητεία θα έχουμε δύο φορέ την ευκαιρία να επιλέξουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο. Στην ε, καταπολέμηση τη ρήπανση τη ατμόσφαιρα, οι δημόσιε συμβάσει αποτελούν όντω ένα σημαντικό κίνητρο για την μετάβαση σε μια κινητικότητα χαμηλών εκπομπών οι αρχές θα πρέπει να δράσουν ε, υποδειγματικά. Και η δική μου κυβέρνηση, η φλαμανδική ε, κυβέρνηση, είναι υπέρ μιας τέτοιας βιώσιμης πολιτικής. Χρειάζεται λοιπόν η μετάβαση αυτή για την ε, καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, αλλά και για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στις πόλεις μας και στις κοινότητές μας και κυρίως στη χώρα μου. Για την, το κόμμα μου, για το NVA, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξουν στην συμφωνία τεχνολογικά ουδέτερε λύσει, όχι μόνο α, οχήματα με μπαταρία και ηλεκτρικά, αλλά υβριδικά με ε, υγροποιημένο αέριο κτλ. Χρειαζόμαστε όλε τι δυνατότητε για να μπορέσουμε να κινηθούμε πραγματικά προ μια κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ συναδελφέ. Και τώρα από την Άλτε το λόγο έχει η κυρία Μιλμπάου Μαραντίκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, θέλω να συγχαρώ καταρχήν τον εισηγητή και όλους τους κοιόδης εισηγητές. Αυτή η πρόταση πρέπει να δώσει δύο βασικά χαρακτηριστικά στον κοινό μας στόχο της μείωσης των εκπομπών στις μεταφορές κατά 20% μέχρι το 2025. Ε, δύο βασικά χαρακτηριστικά, ρεαλισμό και σαφήνεια. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για να ε, σχετικοποιήσουμε τα όσα λέγονται για τον δίζελ. Γιατί μας, ε, το δίζελ ε, μας εμποδίζει να μειώσουμε ε, το, τις εκπομπές, περιμένοντας τις μηδενικές εκπομπές και δημιουργεί μεγάλο κοινωνικό κόστος, διότι ήδη βλέπουμε μείωση στις, στην απασχόληση εξαιτία της κρίσης του δίζελ. Και υπάρχουν εναλλακτικέ που είναι πολύ πιο καθαρές από τον δίζελ. θα πρέπει η μετάβαση να γίνει σταδιακά προς τις μηδενικές εκπομπές. Ε, θα πρέπει να μπορούμε με ρεαλισμό να καθορίσουμε σαφείς στόχους για το μέλλον. Άλλες ε, χώρες, στους οποίους πουλούν οι δικοί μας κατασκευαστές, το έχουν ήδη κάνει. Προβλεψιμότητα και ρεαλισμός ε, θα πρέπει να βοηθήσουν και τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να ε, διοχετεύσουν τις επενδύσεις τους με τρόπο έτσι ώστε να αποδώσουν στο μέλλον. Γι' αυτό το λόγο αυτό το κείμενο πέραν το ότι θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κρίσης της πωλήση, θα βοηθήσει, θα ενθαρρύνει μια βιομηχανική πολιτική προς τα οχήματα μηδενικών εκπομπών. Επίσης, ε, θα επιτρέψει σε κάθε τύπο μεταφοράς να προσφέρει ό,τι μπορεί σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, ε, την κοινωνική αποδοτικότητα και την περιβαλλοντική αποδοτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, η εμφάνιση νέων τύπων πρόσβασης στα οχήματα. Για παράδειγμα, σε ορισμένε ε, χώρες, όπως τη δικιά μου, ο μέσος όρος ηλικίας των αυτοκινήτων από 8 έτη το 2007 πέρασε στα 12,4 το 2017. Το 62% μάλιστα έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών. Και θα φτάσει και μερικέ φορέ στα βαν, στα μικρά επαγγελματικά οχήματα, φτάνει τα 13 έτη. Το να μπλοκάρουμε την ανανέωση του στόλου περιμένοντα τα οχήματα μηδενικών εκπομπών είναι πολύ κακό. Θα ήταν πολύ κακή είδηση και για το περιβάλλον και για την οδική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, ο κύριος, η κυρία Κονέτσινα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Ποιο είναι πραγματικά το αποτέλεσμα αυτό. Υπερβολικές απαιτήσει στους παραγωγούς για τη μείωση των εκπομπών και τίποτα άλλο. Το κείμενο της οδηγίας για την πρόθεση των ε, αποδοτικών οχημάτων ε, θα έπρεπε να οδηγεί σε μια αγορά ελεύθερων, ε, καθαρών οχημάτων, αλλά έχει φτάσει πάρα πολύ αργά και περιλαμβάνει πολλά παραθυράκια. Οι, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να δαπανίζουν δισεκατομμύρια ευρώ για να αναπτύξουν αυτές τις τεχνολογίες, αλλά ποιος θα τις αγοράσει ο κρατικός τομέας ε, δεν είναι έτοιμος ακόμα. Τα κράτη-μέλη μεταθέτουν το φορτίο και το κόστος στους κατασκευαστές. Στην πραγματικότητα δεν θα επιτευχθεί μείωση εκπομπών. Τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς επίσης δεν ήταν ικανοποιητικά. Η, η περίοδος μεταγραφής είναι πάρα πολύ μικρή, δεν είναι ικανοποιητική το Κοινοβούλιο πούλησε το θέμα αυτό πολύ φτηνά. Δεν μπορώ να στηρίξω αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον τελευταίο ομιλητή, είναι η τελευταία φορά, θα σας πω, που προεδρεύω στην Ολομέλη αυτή, αυτή τη θητεία. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την δυνατότητα που μου δώσατε εσείς οι πολλοί και οι λίγοι εδώ σήμερα να είμαι αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια της ιδέας μου προσπάθησα να τιμήσω την θέση αυτή με συμμετοχή, δέσμευση και βούληση να υλοποιήσω τις δεσμεύσεις που είχα αναλάβει όταν ε, προσπάθησα να επαναφέρω τον πλουραλισμό μέσα στο Προεδρείο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας βάθους καρδίας και ε, καλή επιτυχία σε όλους όσοι κατεβαίνουν στις εκλογές για να βελτιώσουν την Ευρώπη προς όφελος όλων των πολιτών της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Για τους ε, πράσινους, ο κύριος Μαρτσελέζη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως έλεγε χθε η Γκρέτα Τόμπερ, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο σπίτι, το σπίτι μας ε, ε, καταραίει. Αυτό έχουμε μπροστά μας μια κλιματική κρίση και χρειάζεται σήμερα, χτες, μια λύση. Ο, ο, κλάδος των οδικών μεταφορών είναι από τους πιο ρηπογόνους. Σύμφωνα, συμφωνούμε σήμερα να βελτιώσουμε την κατάσταση ζητώντας από όλα τα κράτη-μέλη ε, να αντιμετωπίσουν χρησιμοποιήσουν το 20% των οχημάτων με, καθαρότερο τρόπο. Αυτό σίγουρα είναι βελτίωση. Ωστόσο, όπως θύμισε χτες η Γκρέτα Τόμπεργκ, μπροστά στην κρίση δεν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, αλλά ό,τι είναι δυνατό. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια πραγματική επανάσταση στον κλάδο των μεταφορών και της κινητικότητας, μια, μετα, μια επανάσταση στην υγεία και το κλίμα. Για παράδειγμα, στις πόλεις της Ισπανίας, ε, Βαλένθια, Μαδρίτη, γίνεται μία μετάβαση σε μία βιώσιμη μετακίνηση χωρίς καύσιμα, χωρίς ορυκτά καύσιμα. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας, ε, ένας θα έχουμε ένα στόλο ε, λεωφορείων καθαρά 100% ε, χωρίς, ε, ε, χωρίς ε, ορυκτά καύσιμα του χρόνου. Αυτό είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει ολόκληρη η Ευρώπη. Είναι δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σβολικανιά. Ένα λεπτό από Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μεταφορέ στην Ευρώπη θα πρέπει να γίνουν πιο καθαρές και θα χρειαζόμαστε πιο φιλικές προ το περιβάλλον οδού μεταφορά. Ε, και νομίζω ότι είναι σωστό το γεγονό ότι με την οδηγία αυτή θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι οι δημόσιε προμήθειε θα δώσουν το καλό παράδειγμα, κυρίως σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία, γιατί οι δημόσιε μεταφορές αποτελούν 75% των, ε, δημόσιες μάλλον αγορές ε, το από πλευρά των κρατών αποτελούν 75% των συνολικών και έτσι Στη Γερμανία έχουμε πολλά καλά παραδείγματα. Το Βερολίνο μέχρι το 2030 θέλει να είναι χωρίς εκπομπές ε, μέχρι το 2030 και ήδη στην πατρίδα μου έχουμε ηλεκτρικά λεωφορεία, πιο πολύ από ό,τι σε όλη την υπόλοιπη Γερμανία. Όλα αυτά είναι εφικτά λοιπόν και γι' αυτό είναι σημαντικό και τα λεωφορεία με βιοαέριο να αναγνωριστούν για ε, την, ε, τα λεωφορεία αστικά λεωφορεία που καλύπτουν μεγαλύτερε αποστάσει. Και νομίζω λοιπόν ότι κάνουμε ένα πολύ καλό και σημαντικό βήμα με την τρέχουσα νομοθεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα η κυρία Σάλντε Μούζα είναι η επόμενη μιλήτρια για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αντιμετωπίζουμε πολλά κλιματικά προβλήματα και νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Όλοι όσοι παρακολουθούμε και τις εξελίξεις. Και χθες αυτό μας είπε και η Γκρέτα Τούνμπερκ. Έχουμε λοιπόν προβλήματα σε ό,τι αφορά και τις πολιτικές και σε ό,τι αφορά την ε, ρήπανση της ατμόσφαιρας που είναι πολύ φτωχής ποιότητας. Τα καθαρά οχήματα είναι τμήμα τη λύση, θεωρώ, και πραγματικά θα μπορούσαμε να έχουμε θέσει του στόχου σε πιο υψηλό επίπεδο, να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Παρ' όλα αυτά, κάτι κάνουμε τουλάχιστον τώρα θέτουμε δεσμευτικού στόχου για του δήμου και τι κοινότητε σε ό,τι αφορά την πολιτική των δημοσίων συμβάσεων, τι αγορέ, τι δημόσίε των οχημάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν επιλύει το πρόβλημα τη ρήπανση τη ατμόσφαιρα, δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον είναι ένα σημαντικό βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Ελπίζω, ελπίζω το επόμενο κοινοβούλιο να δείξει πιο υψηλό επίπεδο φιλοδοξία από ό,τι και εμεί. Καλωσορίζουμε παρόλα αυτά το γεγονό ότι γίνεται μία βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπούλτς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Okay. Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Χαίρομαι που παρατηρώ πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να στηρίζει ε, αυτή την πρόταση. Θέλω να ξαναευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές για τις επικοδομητικές διαπραγματεύσεις που μας επέτρεψαν να συμπληρώσουμε, να, να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή έγκαιρα πριν διακόψει το Κοινοβούλιο μαζί με, άλλα τα, μαζί με τα άλλα στοιχεία των πακέτων κινητικότητα 1-2-3, η αναθεωρημένη οδηγία θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να μας βοηθήσει να πετύχουμε σημαντικές μειώσεις εκπομπών στον τομέα των μεταφορών, που είναι απαραίτητες προκειμένου να τηρήσουμε τις δεσμεύσει μας με τη Συμφωνία COP21 του Παρισιού η υιοθέτησή της θα αποτελέσει έγκυρη, έγκαιρη συγγνώμη, συνεισφορά στην επίτευξη αυτών των στόχων μέχρι το 2025. Πριν κλείσω, θα ήθελα όμω να κάνω ένα-δύο σχόλια στα όσα είπατε. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το επίπεδο φιλοδοξίας μας. Πράγματι, αυτό το πακέτο, αυτή η πρόταση, είναι φιλόδοξη. Αλλά αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Ακριβώς αυτό ταυτόχρονα είναι και ρεαλιστική και συνάδει με τις προβλέψεις για την αγορά. Να υπογραμμίσουμε ότι η πόλη, η τη σημαντικά δίκτυα δηλαδή πόλεων, ε, τοπικές, ε, η Local Governance for Sustainability, το Συμβούλιο Δήμων και Κοινοτήτων έχουν ε, εκφράσει και στο Κοινοβουλίο και στην Ρωμανική Προεδρία την πλήρη στήριξή του στην πρόταση της Κομισιόν. Οπότε ναι, ε, οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές αρχές είναι έτοιμες. Τα οχήματα με μηδενικές εκπομπές αυτή τη στιγμή στηρίζονται σε... Ε, ε, είναι, έχουν ψηλή τιμή, αλλά αν το κόστος αυτό διαρρεθεί με το χρόνο ζωής τους, μειώνεται και θα μειωθεί ακόμα περισσότερο μέχρι να εφαρμοστεί η Οδηγεί αυτή, πολύ δε περισσότερο, που οι οικονομίες κλίμακος θα ρίξουν ακόμα περισσότερο το κόστος. Η οικονομική στήριξη είναι απαραίτητη, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουμε και υπάρχοντα ε, ε χρηματοδοτικά όργανα όπως το Connecting Europe, Facility, ε, το EFSI κλπ. Να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει ένα κονδύλιο ακόμα και για τα ηλεκτρικά λεωφορεία, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται από πολλές ε, ευρωπαϊκές πόλεις. Οπότε είναι σημαντική η σαφής στόχη για τις κρατικές προμήθειες και θα διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία. Ένα σχόλιο τώρα σε ό,τι αφορά μάλλον κάποιες περισσότερες πληροφορίες για την αυτοκινητοβιομηχανία. Τον Ιούνιο του 2018 μια ομάδα μεγάλων αυτοκινητοβιο... αυτοκινητοβιομηχανιών, Solaris, Skoda, Volkswagen, Ursus κλπ. Έστειλαν μια ανοιχτή επιστολή στο Συμβούλιο και ζητούσαν περισσότερα φιλόδοξους στόχους από αυτούς που πρότεινε η Κομισιόν και επιβεβαίωναν ότι είναι έτοιμες να ανταποκριθούν. Οπότε ενθαρρυνόμαστε σε αυτή μας την, ε, σε αυτήν την κατεύθυνση που κινούμαστε και από τις δύο πλευρές, και από τους αγοραστές και από τους πολιτές. Επίσης να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε. Πολλέ μεγάλες πόλεις ήδη έχουν ξεπεράσει τους στόχου σε ό,τι αφορά στις, ε, ε, στις ε, δεσμεύσεις τους. Ο στόχο τη οδηγία είναι να ενθαρρύνει και άλλε πόλεις να ακολουθήσουν αυτό το καλό παράδειγμα, αναγνωρίζοντας ότι πολλές μικρές και μεσαίε πόλεις ενδεχομένω δεν είναι ακόμα έτοιμε, δεν έχουν επαρκή τεχνογνωσία ή πόρου όπω το Άμστερνταμ ή το Παρίσι. Είμαστε όμω έτοιμοι να τις βοηθήσουμε για να διαπραγματευτούν από κοινού καλύτερες τιμές με την αυτοκινητοβιομηχανία. Οπότε αναμένω να υιοθετηθεί η έκθεση ε, του κύριου Ξιπ αύριο. Αυτό το θέμα, αυτό το κείμενο αποδεικνύει ότι αναγνωρίζουμε τη σαφή ανάγκη και ότι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά ωφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Yes, Ευχαριστούμε, κυρία Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα θετικά σας λόγια. Οπότε τώρα θα ακούσουμε τον εισηγητή μας, τον κύριο Ξύπα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο ηλεκτρισμός ως πηγή ενέργειας είναι πράγματι πολύ αποτελεσματική πηγή για τα αυτοκίνητα. Είναι βέβαια ακριβώς, ακριβή πηγή. Επίσης γνωρίζουμε ότι στηρίζοντας την ανάπτυξη του τομέα αυτού, δηλαδή των καθαρών οχημάτων, σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές και στην παραγωγή, στην κατασκευή ε, οχημάτων. Πώς θα πείσουμε λοιπόν τον κόσμο εφόσον θα έχουμε πιο καθαρό αέρα, ατμόσφαιρα. Τα καθαρά οχήματα βοηθούν να έχουμε πιο καθαρή ατμόσφαιρα, άρα αυτό ακριβώς που θέλει ο κόσμος και ζητά. Και έχω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπάρχει ένας καθηγητής σε μια πολωνική πόλη που του αρέσει να τρέχει. Και μετά από πολλά χρόνια που έτρεχε είπε «Ξέρω ότι έχω κάνει κάτι στραβό, κάτι λάθος, γιατί τώρα έχω πρόβλημα με τα πνευμόνια μου. Αυτό δείχνει πόσο πολλοί είναι οι πολίτες που τελικά έχουν προβλήματα στην αναπνοή, πεθαίνουν πρόωρα εξαιτίας της ρήπανσης της ατμόσφαιρας. Όλο περισσότερες πόλεις βλέπουν τις αρχές τους να αποφασίζουν να περιορίζουν την πρόσβαση των οχημάτων στο κέντρο των πόλεων αυτών. Και τα μόνα οχήματα τα οποία επιτρέπονται είναι τα ηλεκτρικά. Και αντιλαμβάνομαι αυτό που είπε κάποιος νωρίτερα εδώ, ότι σίγουρα επιβάλλονται περιορισμοί από τις χώρες μέλη, από τις τοπικές αρχές, σε μερικές περιπτώσεις, αλλά δεδομένων των επαφών που έχω με την τοπική αυτοδιοίκηση σε περιφέρειες, πόλεις, δήμους κτλ. Πρώτα γίνονται διαβουλεύσεις και μετά λαμβάνονται αποφάσεις. Και βλέπω ότι ο κόσμος τελικά θέλει να δεχτεί τον ευρύτερο ορισμό για οχήματα μηδενικών εκπομπών, καθαρά οχήματα που κυκλοφορούν με μεθάνιο, οτιδήποτε άλλο πρέπει να προσαρμόσουμε επίσης τα οχήματα που ήδη βρίσκονται στην αγορά. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία έχουμε αναπτύξει στις διαβουλεύσεις που έχουμε τους κοινωνικούς εταίρους και με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους, κυρίως τις τοπικές αρχές, γιατί μας λένε τι περιμένουν να περιλαμβάνει η νομοθεσία αυτή προκειμένου να γίνει αποδεκτή. Εννοείται ότι πρόκειται για ένα συμβιβασμό μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων του Κοινοβουλίου, ε, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε θέλω να εκφράσω εδώ τις ευχαριστίες μου σε όσους συμμετείχαν στην εκπόνηση αυτού του κειμένου. Αυτό που πρέπει επίσης να γνωρίζετε είναι ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια μετά το 2020 θα στηρίξουν τους στόχους της οδηγίας. Και είναι και αυτό ένα κίνητρο για εκείνους που θέλουν να εμπλακούν στην υλοποίηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τη συνεργασία σας, όλους σας, για τη συνεργασία σας όχι μόνο στην ε, οδηγία αυτή ε, και σας, γιατί όλοι μαζί συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε κάτι. Δεν συμφωνούμε πάντα όλοι σε όλα, αλλά πιστεύουμε όλοι ότι κάνουμε κάτι καλό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Η ψηφοφορία για το θέμα αυτό θα λάβει χώρα αύριο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μπούλτς για την παρουσία της εδώ. Καλό σας βράδυ. Και καλωσορίζω εδώ την κυρία Γιούροβα, την Επίτροπο Γιούροβα και θα συζητήσουμε τώρα μαζί της την έκθεση του κυρίου Ταντέου Σβιεφκά πρόκειται για την χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου. Η έκθεση του κ. Ζιέφκα. Έχετε το λόγο, κ. Ζιέφκα. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να απευθυνθώ σε εσά, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, βλέπουμε ότι η θητεία ολοκληρώνεται, αλλά υπάρχουν ακόμα αρκετά σημαντικά θέματα τα οποία και πρέπει να εγκρίνουμε. Η ευρωπαϊκή αγορά, οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη περιμένουν και θα ήθελα ευθύ εξ αρχή ε, να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο, την κυρία Γιούροβα. Ε, επίσης, να ευχαριστήσω την ομάδα της γιατί ε, έκαναν ε, πάρα πολύ καλή δουλειά, ε, κατέθεσαν μια θαυμάσια πρόταση και έτσι περιόρισαν και το χρονικό διάστημα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Κατέστη λοιπόν δυνατόν να διεξάγουμε τις διαπραγματεύσεις στον τριμερή διάλογο με απόλυτη ηρεμία και ησυχία. Ευχαριστώ τους και τις εισηγήτριες, τους συναδέλφους μάλλον, που ήταν σκιώδη εισηγητές. Περί πρόκειται, πρόκειται για το εταιρικό δίκαιο που είναι πολύ σημαντικό για την κοινή αγορά. Και πρόκειται κατ' ουσίαν και για ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί την κοινωνία, την ψηφιοποίηση. Η νέα οδηγία δίνει νέες δυνατότητες για την καταχώρηση των επιχειρήσεων, όπου ε, μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί τις ε, ψηφιακές ε, τεχνολογίες, συγκεκριμένα το διαδίκτυο. Είναι βέβαια λίγο περίεργο το ότι μόνο στο τέλος της θητείας συζητάμε για την ψηφιοποίηση σε σχέση με τα δικά μας τα θέματα για την κοινωνία της πληροφορίας. Μιλάμε αρκετό καιρό, αλλά τώρα αυτό που ενδιαφέρει είναι το τι προσδοκούν οι εταιρείε από εμάς. Κυρίες και κύριοι, ένα πράγμα είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ο στόχος που έχουμε είναι η βελτίωση, η διευκόλυνση της ζωής των εταιριών σε αυτό το θέμα της καταχώρησής τους. Πρόκειται για έγγραφα, παραστατικά, το πώς ε, διαβιβάζονται, ε, το πώς γίνεται ο συντονισμός ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, βέβαια υπάρχουν ήδη αυτές οι δυνατότητες, αλλά η όλη διαδικασία ήταν χρονοβόρα και δαπανηρή. Και υπάρχει και μια ανασφάλεια σχετικά με το πώς γίνεται η καταχώρηση σε ένα άλλο κράτος μέλος. Έτσι λοιπόν, πρόκυψε το εξής. Οι δυνατότητες στην αγορά εξαφανίστηκαν ή εξαφανίζονται πριν καν δραστηριοποιηθεί μια εταιρεία. Μια εταιρεία ή δεν υφίστατο καθόλου ή ήταν αναγκασμένη να παραιτηθεί από συμβάσεις γιατί ο χρόνος για καταχώρηση ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Τώρα λοιπόν με αυτή την πρόταση περιορίζουμε το χρόνο καταχώρησης. Η ψηφιακή καταχώρηση πρέπει να, μπορεί να γίνεται από 5 μέχρι το πολύ 10 ημέρες. Βεβαίως ε, πρέπει να εκπληρώνονται όλες οι υποχρεώσεις, ε, ε, πρέπει να κατατίθενται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και βεβαίως στην οδηγία εκφράσαμε κάποιες επιφυλάξεις για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου απάτης κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με τα θέματα που συζητάμε. Κυρίες και κύριοι, πολύ συγκεκριμένα, για ποιες επιχειρήσεις πρόκειται, έχω στοιχεία που δείχνουν ότι έχουμε περίπου 24 εκατομμύρια εταιρείες στην Ευρώπη και περίπου το 80% εξ αυτών είναι κεφαλαιακές εταιρείες και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 não estava garantido à partida. Porquê? Para nós, Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ισχύουν αυστηρέ προδιαγραφέ κατά των απατών, όταν δηλαδή τα κράτη δίνουν τη δυνατότητα στι εταιρείε να συστήνονται με ένα απλό πάτημα του ποντικού. Εμεί δεν θέλουμε να υπάρχουν εικονικέ εταιρείε, ούτε να προάγουμε επιχειρηματικά μοντέλα που ορίζονται ω το Delaware τη Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε πάρα πολύ πολύ τον κύριο Συγητή, την κυρία Επίτροπο, συγχαρητήρια στην διαπραγματευτική ομάδα, στην Σκιώδη Συγήτρια. Το αποτέλεσμα προβλέπει το εξή. Ο δεσμευτικό έλεγχο τη ταυτότητα των ανθρώπων που θέλουν να συστήσουν την εταιρεία ε, τα κράτη-μέλη παρά την πλήρη ψηφιοποίηση για λόγους δημοσίου δικαίου μπορούν να καλέσουν αυτά τα άτομα να παρουσιαστούν στην αρμόδια υπηρεσία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε η επιγραμμική καταχώρηση να μην γίνει ένα εργαλείο για εικονικές εταιρείε. Νέε λοιπόν προϋποθέσεις, καλύτερη πληροφόρηση, αυτά θα πρέπει να φαίνονται από τα μελλοντικά λογιστικά στοιχεία για να μπορεί να λειτουργεί και το σύστημα BRIS. Αυτό που έχει η σημασία είναι ότι στο μέλλον σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εισαχθούν κανόνες έτσι ώστε να αποκλείονται κάποια στελέχη από τις εταιρείε, οι απαταιώνες δεν θα πρέπει να μπορούν να εξαπατούν ε, άλλα κράτη-μέλη. Οι επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να μπορούν να εκμεταλλεύονται την ψηφιοποίηση, αλλά η Ευρώπη δεν θα μπορεί να γίνει ένα σούπερ μάρκετ ε, ψηφιοποίηση με τις αυστηρές προδιαγραφές και με τον έλεγχο της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Τα κράτη-μέλη θα μεριμνούν έτσι ώστε να μην προκύπτει κατάχρηση του εταιρικού δικαίου. Συγχαρητήρια λοιπόν για το σπριντάρισμα. Θα το το χαρακτηρίσω αν μου επιτρέπετε, το οποίο κατορθώσαμε έστω και στο τέλος της θητείας αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε. Επόμενος πακέτ εκ μέρου του ECR. Έχετε το λόγο. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στην Φλάνδρα οι μικρομεσές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν και τη σποδηλική στήλη της οικονομίας. Ε, ζούνε χιλιάδες και χιλιάδες οικογένειες από αυτές. Τώρα μιλάμε για την ψηφοποίησή τους. Και μιλάμε και για το δίκαιο που όντω πρέπει να συνοδεύει αυτή την ε, ψηφιοποίηση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και για να συμβεί αυτό πρέπει οι χώρες μέλη να φροντίσουν η ψηφιοποίηση αυτή να γίνει όσο γίνεται πιο απλά. Οι δυνατότητες μιας επιχειρίας να οργανωθεί ψηφιακά δεν πρέπει να επιτρέπει κανένα περιθώριο απάτης. δεν ε, θα πρέπει να υπάρχουν παραθυράκια ώστε να μπορεί να γίνεται νομιμοποίηση, για παράδειγμα, παράνομου χρήματος. Πρέπει να βρεθούν τα μέσα εκείνα τα οποία θα εγγυηθούν για την ασφάλεια, μέσα για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση ή οτιδήποτε άλλο για την καταχώρηση στο Μητρό. Όντω, για τι επιχειρήσει τα πράγματα πρέπει να γίνονται πιο εύκολα, πιο απλά. Πρώτα απ' όλα γιατί έτσι εξοικονομούν χρήματα αλλά και γιατί θα μπορέσουν να δημιουργηθούν και περισσότερες επιχειρήσεις. Και αυτό σίγουρα θα είναι θετικό εφόσον θα γίνεται ηλεκτρονικά η καταχώρησή τους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Σφίρσκα για να κλείσει τη συζήτηση, προηγουμένως η Επίτροπος έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις σας όλους και πράγματι σας ενθαρρύνω να υπερψηφίσετε το κείμενο αυτό, αυτή την πρόταση. Με την νομοθετική αυτή πρόταση, όντως, καλούμε τις μικρομεσαίες και γενικά τις επιχειρήσεις στον 21ο αιώνα. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Κάνουμε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Επίσης, μπορούμε τώρα να επικεντρώσουμε και τις προσπάθειές μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η υλοποίηση ε, θα γίνει εφικτή και στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για τις τελευταίες του σκέψεις από αυτού και συγχαρητήρια και για το έργο σας έτσι κι Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την Επίτροπο και όλους τους συναδέρφους για τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται έτσι μια μεγάλη διαδικασία συνεργασίας κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Για μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συνομοθέτης, είναι προφανές ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις αποτελούνται από ανθρώπους με κυριότητα, οι οποίοι δεν θα προβούν σε απάτες. Προτείνουμε λοιπόν καλές λύσεις για να διευκολύνουμε την καθημερινότητά τους. Η καθημερινότητα είναι ψηφιακή έτσι καλλιώς σήμερα. Απάτες πάντα συνέβαιναν και πάντα θα συμβαίνουν. Και στην κλασική καταχώρηση δεν βλέπω γιατί τώρα να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για απάτες. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στις εργασίες μας και συνεισέφεραν επενδύοντας χρόνο και έργο για να ετοιμαστεί αυτή η νομοθετική πρόταση. Και προς το Συμβούλιο θέλω να πω ότι δεν πρέπει να αργήσουμε να εφαρμόσουμε την οδηγία αυτή. Οι πολίτες μας περιμένουν ανυπόμονα αυτό το νομικό μέσο που είναι τόσο σύγχρονο και ελπίζω αυτό να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε εδώ τη συζήτηση. Αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία για την έκθεση αυτή. Στη συνέχεια, αγαπητοί συνάδελφοι, στην ημερησία διάταξη έχουμε την έκθεση της κυρίας Εύελιν Ρέγκνερ, διασυνοριακές μετατροπέ συγχωνεύσει και διασπάσεις. Καταρχήν, θα ακούσουμε την εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Αυτό το οποίο καταφέραμε εδώ είναι ένα ορόσημο. Η οδηγία είναι περίπλοκη, είναι πολύ διευρυμένη, έχει σχέση και μπορεί να συγκριθεί με την οδηγία περί προστασίας δεδομένων, παραδείγματο χάρη, σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορέσαμε να συνδυάσουμε την εντολή των δύο θεσμών και να επεξεργαστούμε ένα κοινό κείμενο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους, την Επιτροπή, ε, την Επίτροπο, τους και οδησηγητές, αλλά και το Συμβούλιο. Έχουμε λοιπόν ένα νέο ε, νόμο ο οποίος ε, προβλέπει και ρυθμίζει την κινητικότητα των επιχειρήσεων και εισάγει μια ενιαία διαδικασία για τις ε, συγχωνεύσεις και τις διασπάσεις των εταιριών. Ναι, πράγματι όλες οι εταιρείε έχουν το δικαίωμα να μετεγκαθίστανται σε μια άλλη χώρα. Εγώ Προέρχομαι από τα συνδικάτα και θεωρώ ότι τα οι εταιρείε θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο που αυτό το δικαίωμα ποτέ δεν απέτυχε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Γι' αυτό λοιπόν ε, ισχύει η νομολογία, αλλά η νομολογία ήταν πέρα από τους νόμους και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στο να δημιουργηθούν εικονικές εταιρείε. Γι' αυτό εμένα αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια ισορροπία. Οι εταιρείε μπορούν να ασκούν ε, το δικαίωμά τους, αλλά όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, κυρίως οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να είναι σωστά προστατευόμενοι. Μπορέσαμε να βρούμε έναν καλό κοινό παρονομαστή. Οι βασικέ προποθέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμφανίζονται σε αυτή τη νέα οδηγία. Καλύτερη προστασία των εργαζομένων όταν τα κράτη-μέλη μετακινούνται σε άλλο κράτο μέλο. Και επίση ε, και μια δεσμευτική ρήτρα κατά των καταχρήσεων ε, για να μπορούμε ακριβώ να αποφύγουμε αυτέ τι εικονικέ εταιρείε. Ε, το θέμα του προσωπικού με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εισακούνται, να ενημερώνονται όταν πρόκειται για την ύπαρξή τους και για, ε, και για την εργασία τους. Η σωστή ενημέρωση των εργαζομένων επιτρέπει στο μέλλον να είναι δικαίωμα η ενημέρωση των εργαζομένων για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Να υπάρχει δεσμευτική, υποχρεωτική, να υπάρχουν υποχρεωτικά διαβουλεύσεις και επιπλέον εισάγονται και νέα ε, δικαιώματα για τους εργαζόμενους ε, όταν μια χώρα μετεγκαθίσταται. Ε, οι εργαζόμενοι στο μέλλον θα έχουν μια εκτενή έκθεση στα χέρια τους για το μέλλον των θέσεων απασχόλησής τους. Θα ερωτώνται για τη μετεγκατάσταση, θα μπορούν έγκαιρα να τοποθετούνται και για πρώτη φορά αποκτούν το δικαίωμα να ζητούν αιτιολογημένη άποψη από την διοίκηση. Επίσης, καθίσατε σαφές ότι οι εθνικοί κανόνες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους ε, τις, ε, τους ενωσιακούς ε, κανόνες και επίσης το ότι τα εργοστασιακά συμβούλια θα πρέπει να έχουν επαρκείς πόρους για να μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Το θέμα του συναποφασίζει, βελτιώνεται με την πρόταση της Επιτροπής και εδώ προβλέπεται προστασία τεσσάρων ετών και αυτό ισχύει για ε, ορισμένα, για όλα τα κρατημέλη, κάτω βέβαια από ορισμένε προποθέσει. Ο δεύτερο τομέα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ απορρέει από την εργασία που έκανα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ε, φορολογικά σκάνδαλα, τα LuxLeaks, ε, τα Panama Papers και πολλά συναφή ε, όσον αφορά την απόσπωση των εργαζομένων, κυρίω στον τομέα των μεταφορών. Εκεί υπάρχουν πολύ συχνά καταχρήσει μέσω των εικονικών εταιριών. Το εταιρικό δίκαιο συστηματικά είναι αντικείμενο καταχρήσεων για να βρουν ενδιαφερόμενοι ζητούμενοι τις καλύτερες συνθήκες, ε, συνήθως εις βάρος στην πλάτη των εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ υπερήφανη για μια δεσμευτική ρήτρα κατά των καταχρήσεων που προβλέπεται πλέον η αρμόδια υπηρεσία στην οποία το δικαστήριο πρέπει να απευθυνθεί. Εάν η αρμόδια υπηρεσία υποπτεύεται ότι υπάρχει κατάχρηση, πρέπει να εξετάσει τις τρεις υποχρεωτικές διαδικασίες ε, κατά πόσον πράγματι τηρήθηκαν τα εθνικά και τα ε, ενωσιακά δικαιώματα, μήπως έγιναν κάποιες προσπάθειες παράκαμψή τους ή μήπως υπάρχουν άλλοι εγκληματικοί στόχοι. Εάν διαπιστωθεί ότι ισχύει κάτι από όλα αυτά, τότε δεν θα δίδεται η άδεια σε μία εταιρεία. Εάν λοιπόν μία εταιρεία τελήσει, να παρακάμψει δικαιώματα ή να συστήσει παράνομα εικονικές εταιρείες, τότε η μετεγκατάσταση απαγορεύεται. εικονικες είναι λοιπόν η ρήτρα που ισχύει και για συγχωνεύσεις και για διαιρέσεις εταιριών, αυτή η συγκεκριμένη ε, οδηγία παίρνει σάρκα και οστά. Εάν μετά την αναδιάρθρωση προκύψουν ύποπτες εξελίξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα. Με την κινητικότητα των εταιριών δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πλέον καταχρήσεις και εικονικές εταιρείε. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα εκτεταμένο πακέτο, μία δέσμη μέτρων που μου επιτρέπει να ευχαριστήσω όλους τους και τον κύριο Ντεγκράντε και τον Πασκάλ Ντιγόν, οι οποίοι όλοι προσπάθησαν αυτή την ε, εκτεταμένη δέσμη μέτρων επιτέλους να την ε, καταστήσουν σε κάτι το απόλυτα συγκεκριμένο. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιούροβα έχει το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Θα ξεκινήσω την ομιλία μου με συγκίνηση, γιατί είναι η τελευταία ολομέλεια για μένα στη θητή αυτή. Συμμετείχα σε τόσες ε, πολλές ε, την τελευταία πενταετία και πρέπει να πω ότι εργαστήκαμε για πάρα πολλά θέματα και με την κυρία Ρέγνερ και με τον κύριο Ντεγκράντες και πάντοτε αισθανόμουν ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη η συνέργεια πολιτικής βούλησης, ε, λογικής ε, και κατανόησης. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα, αυτό το πακέτο εταιρικού δικαίου, ε, που είναι πολύ πολύπλοκο, αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα. Και Πολλοί δεν πίστευαν ότι θα τα καταφέρναμε να το ολοκληρώσουμε. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέλος μιας πολύ δύσκολης αλλά επιτυχούς διαδικασίας. Η Ευρωπαϊκή Αγορά προσφέρει πολλές ευκαιρίες στις εταιρείε ε, να αναπτυχθούν. Όμω πολύ συχνά οι εταιρείε ε, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ωφέλη στην πράξη. Η πρόταση τη Κομισιόν απάντησε ε, σε αίτημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα συνδικάτα και τι οργανώσει των επιχειρήσεων για νέου κανόνε στον τομέα αυτό. Και θέλω να ευχαριστήσω την συγγήτρια, την κυρία Ρέγνερ ε, και τι αντίστοιχε προεδρίε του Συμβουλίου για την υποκριτική του προσέγγιση και την αποτελεσματική του δουλειά σε αυτή την ιδιαίτερα πολύπλοκη και σημαντική σημαντική πρόταση. Χαίρομαι πολύ που το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρήκαν ένα ρεαλιστικό και καλό συμβιβασμό που θα βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους υπαλλήλους. Η οδηγία θα βοηθήσει τις εταιρείε ε, να μετακατασταθούν και να οργανωθούν στην ενιαία αγορά, ενώ θα παρέχει τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες για τους ε, ενδιαφερομένους και τους υπαλλήλους η Κομισιόν. Καλωσορίζει τον ε, υποχρεωτικό χαρακτήρα των μέτρων κατά της κατάχρησης. Ήταν ένα σημαντικό θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για πολλά από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Κομισιόν καλωσορίζει επίσης τις διατάξεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπου περιλαμβάνονται πολλά από τα θέματα που τέθηκαν στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το κατόφλι των τεσσάρων πέπτων για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ε, και στις ε, τρεις διασυνοριακές πράξεις. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας αυτών των διαπραγματεύσεων και οι διατάξεις προστασία της διαπραγματευόμενης λύσης, ε, αν υπάρχουν και μετέπειτα πράξεις, ε, παρέχουν ένα πλήρες πακέτο ασφαλιστικών δικλείδων. Επιπρόσθετα, το νέο άρθρο για την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών και τη διαβούλευση τονίζει και τα δικαιώματα των υπαλλήλων να έχουν λόγο σε μια διασυνοριακή διαδικασία. Και αυτό ήταν ουσιαστικό για το Κοινοβούλιο. Ε, θυμόμαστε τι αποκλίνουσε θέσει που υπήρχαν όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσει. Και η Κομισιόν θα ήθελε να συγχαρεί του συνομοθέτε για τι λύσει ε, που βρέθηκαν ε, για ε, τον συμβιβασμό που αποτελεί ένα καλό βήμα προς τα μπρος σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Παρέχει εύρωστους και δίκαιους κανόνες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ε, που συμμετέχουν στις συνοριακές διαδικασίες, ενώ δεν είναι πολύ βαριά διαδικασία στην πράξη. Επομένως, η Κομισιόν μπορεί να υποστηρίξει πλήρως το συμβιβασμό και ανυπομονή για την αυριανή ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της ΕΚΟΝ, ο κύριος Λούντβικσον, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ήμουν συντάκτης γνωμοδότησης από πλευράς της Οικονομικής Επιτροπής και ετοίμασα την γνωμοδότησή μου που λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ασφαλείς κανόνες οι οποίοι να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μετακινούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις επιχειρήσεις που εργάζονται σοβαρά. Συγχρόνως όμως χρειαζόμαστε και κανόνες που θα μας επιτρέψουν να καταπολεμήσουμε το dumping ε, στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Πρέπει να αποφύγουμε απλώς και μόνο ε, ο στόχος της μετακόμισης να είναι να αποφεύγονται οι κοινωνικοί κανόνες, δηλαδή να μην σεβόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ την εισηγήτρια την κυρία Ρέγνερ και όλους τους σκιώδεις εισηγητέ και όσους γνωμοδότησαν για την καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας και με το Συμβούλιο. Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν τώρα περισσότερες δυνατότητες για ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα στην εσωτερική αγορά. Συγχρόνω, οι νέοι κανόνες προσφέρουν και μία ενισχυμένη ασφάλεια τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους μετόχους των επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό αύριο να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας και είναι επίσης σημαντικό να έχουμε ασφαλείς κανόνες όταν πρόκειται για τα δικαιώματα των επιχειρήσεων μέσα στην εσωτερική αγορά. Συγχρόνως όμως να αποφύγουμε κάθε κατάχρηση, κάθε απάτη είναι πολύ σημαντικό γιατί αλλιώς θα υπονομευθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην εσωτερική αγορά. Μέσα από το κείμενο αυτό είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε περισσότερη δικαιοσύνη στην ενιαία αγορά. Είναι μια δικαιοσύνη η οποία θα επιτευχθεί εάν πάψουν να υπάρχουν εικονικές επιχειρήσεις. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ε, ξεκινάμε με τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Δεγκράντες Πασκουάλ πρώτα απ' όλα εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Γιούροβα. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ το Συμβούλιο για το έργο του. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια και φίλη μου, αν και αντίπαλος πολλές φορές, την κυρία Ρέγνερ. Εμείς στο ΕΛΚ Στηρίξαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την οδηγία, γιατί ο κύριο στόχο είναι να διευκολύνεται η ζωή των επιχειρήσεων, των μικρομισών κυρίω, και να μπορούν ελεύθερα να μετακινούνται μέσα στην Ευρώπη. Θέλουμε ένα νομικό πλαίσιο μέσα σε ένα κόσμο όλο και πιο περίπλοκο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τους εργαζόμενους, τους μετόχους κλπ. Και γι' αυτό οι νέες εναρμονημένες διαδικασίες περιλαμβάνουν και τις ρήτρες ασφάλειας για να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τα δικαιώματα όλων αυτών. Κυρίε και κύριοι, έπρεπε να δώσουμε μια απάντηση μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ελευθερία εγκατάσταση. Βάσει του άρθρου 49 τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί πάντα υποστηρίζαμε ότι επιχειρήσει οι οποίε εγκαθίστανται σε μια χώρα μέρο έχουν το δικαίωμα και την ελευθερία να μπορούν να μεταφέρουν την έδρα του σε άλλη χωρί να χάνουν τη νομική του προσωπικότητα. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μερικές φορές ακόμα και χωρίς οικονομική δραστηριότητα στη νέα χώρα. Θεωρούμε όμως σημαντικό, όπως και η Συγκίτροπος και το Συμβούλιο, να βάλουμε και μία ρήτρα κατά των καταχρήσεων. Όταν γίνονται τέτοιες διασυνοριακές μετακινήσεις πρέπει να αποφεύγουμε απάτες και κατεχρήσεις του συστήματος. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προσωπικά, όπως ξέρει και η συγγήτρια, υπογράμμισα πάρα πολύ ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δικαιολογούνται. Δηλαδή, αν έχουν πάρει ε, κρατικές επιδοτήσεις, αν έχουν οικονομική ενίσχυση. Δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα, να υποφελούνται δηλαδή από το σύστημα και να αφήνουν ξεκρέμαστους και τους εργαζόμενους. Αυτό θέλουμε και στην Ισπανία. Εμείς επίσης θέλουμε ex post έλεγχο της μετακίνησης για να επαληθεύουμε ότι δεν υπάρχει καμία πάτη και να επικυρώνεται η δραστηριότητα αυτή μόνο εφόσον υπάρχει κατάλληλη εγγύηση για όλους. Το αποτέλεσμα πιστεύω ότι είναι θετικό. Υπάρχει ελευθερία μετακίνησης που ήταν πάντα η προτεραιότητά μας γιατί πιστεύουμε σε μια ενωμένη Ευρώπη χωρίς σύνορα. Αυτό είναι η προτεραιότητά μας και αυτή είναι και η ευθύνη μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τεγκράντες Πασκουάλ. Τώρα ε, για τους σοσιαλιστές ο Μικαέλ Ντέτζεν. Δύο λεπτά. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη Κύριε Επίτροπε, με την αυρινή ψηφοφορία ε, δίνουμε τέλος σε μια παράδεκτη κατάσταση όπου οι εταιρείε θα μπορούσαν να μετακινηθούν σε μια άλλη χώρα χωρίς να τηρούν τους κανόνες. Χωρίς κανόνες λοιπόν ήταν δυνατόν να αναζητήσει κανείς ε, βραχυπρόθεσμα κέρδος και να εγκασταθεί στη χώρα με τους χαμηλότερους μισθούς και τους λιγότερους φόρους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κανόνες οι οποίοι θα προστατεύουν τους εργαζόμενους σε περίπτωση αναδιάρθρωσης. Η προστασία προστασία στα δικαιώματα ενημέρωση και διαβουλεύσεων. Η προστασία είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στη συνάδελφό μου την κυρία Ρίγνα ε, για την επιτυχία που σημείωσε παρά τις δυσκολίες. Η πρώτη επιτυχία της είναι ότι πλέον από μια χαόδη κατάσταση περνάμε σε μια ρυθμιζόμενη ε, η διοίκηση για πρώτη φορά είναι υποχρεωμένη να καταθέτει στο προσωπικό ένα, μια λεπτομερή έκθεση ε, σχετικά με την αναδιάρθρωση της εταιρεία ε, μία ρήτρα κατά των καταχρήσεων θα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να ελέγχουν τα αίτια της αναδιάρθρωσης. Καλό και αυτό. Έτσι λοιπόν ε, η ε, εξελίξει αυτές και τα φαινόμενα των εικονικών εταιριών μπορούν να αποφευχθούν. Τα κράτη-μέλη βέβαια δεν ήθελαν να κάνουν άλλο ένα μεγαλύτερο βήμα, έχασαν αυτή την ευκαιρία. Αλλά δεν ήταν η Ευρώπη, δεν ήταν αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν οι κυβερνήσει των κρατών μελών που είχαν παρεμποδίσει, που παρεμπόδισαν την καλύτερη προστασία των εργαζομένων. Το Κοινοβούλιο βρήκε καλέ συμβαστικέ προτάσει. Οι προτάσει αυτέ δείχνουν Λοιπόν, το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και στο θέμα της συναπόφασης. Βλέπουμε να υπάρχει μια πλήρης αντίφαση ανάμεσα στα συνδικαλιστικές ελευθερίες και στα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. Το κείμενο για το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο είναι η καλή αρχή για ένα σύστημα κανόνων. Εγώ θα υπερψηφίσω το κείμενο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι επιγόντως απαραίτητο να υπάρχει μια οδηγία πλαίσιο για τη συναπόφαση στην Ευρώπη. Επειδή είναι η τελευταία μου ομιλία στο Κοινοβούλιο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και τους συναδέλφους μου για το ότι μου έδωσαν τη δυνατότητα να εργαστώ και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τέτσερ και καλή τύχη. Ο κύριος Σίτερβαν τώρα για την ΚΟΕ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ του συζητητέ που αγωνίστηκαν ε, κατά τη ε, φοροδιαφυγή ε, και υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δυστυχώ για άλλη μια φορά διαπιστώνω ότι ένα πολύ καλό κείμενο του Κοινοβουλίου νοθεύτηκε στον τριμερή διάλογο. Αυτό το οφείλουμε στο Συμβούλιο που δεν είναι παρόν. Υπάρχουν νέοι κανόνε για το δικαίωμα εγκατάσταση σε μια ευρωπαϊκή χώρα, σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τους νέους κανόνες δυσχεραίνεται η ε, άσκηση δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ε, εμείς θέλαμε να αποφύγουμε τις εικονικές εταιρείε, ε, να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή. Αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη κοινωτικότητα, καλό αυτό, όμως ε, χάνονται τα δικαιώματα των πολιτών, γίνεται κοινωνικό ντάμπινγκ, γι' αυτό λοιπόν εμείς ως αριστεροί, όπως και ο συνάδελφος, ζητάμε μια οδηγία πλαίσιο για τη συναπόφαση, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι ο κύριος Βόμποντα απουσιάζει, επομένως το λόγο έχει ο κύριος Ράντεφ. Έχετε μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που σήμερα συζητάμε αυτό το νομοθετική πράξη που αποτελεί μέρος του εταιρικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ρέγνερ αλλά και την Κομισιόν γιατί άκουσε την εκκλησή μας για διασυνοριακή εναρμόνιση σε περίπτωση των μετατροπών συγχωνεύσεων και διασπάσεων. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο κύριος σκοπός είναι να διευκολύνουμε τις εταιρείες και κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όταν προβαίνουν σε μετατροπές, ε, συγχωνεύσεις και διασπάσεις διασυνοριακά. Η οδηγία αυτή θα διευκολύνει την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε μεγάλο βαθμό. Ο έλεγχος καταλληλότητας, πιστεύω, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υποχρεωτικά μέτρα κατά της κατάχρησης θα επιτρέψουν στις εθνικές αρχές να σταματήσουν ε, κάποιες τέτοιες πράξεις όταν ε, έχουν ε, απατηλό σκοπό. Εδώ έχουμε διασφαλίσει τα νόμιμα συμφέροντα των πιστωτών, των μετόχων και των εργαζομένων. Οι εργαζομένοι θα πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα για τις συνέπειες των διαδικασιών αυτών και τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας και όσων δεν έχουν δικαίωμα ψήφου θα προστατεύονται. Ταυτόχρονα οι πιστωτές θα έχουν ε, ξεκάθαρες ε, και αξιόπιστες εγγύησεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ράντεφ. Τώρα έχουμε ολοκληρώσει τον κατάλογο των ομιλητών και δεν υπάρχει κάποιος ομιλητής για τη διαδικασία Catch the Eye. Επομένως θα δώσω τον επίτροπο στην κυρία Γιούροβα. Αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, παρεμβάσεις σας για τα θετικά σας σχόλια. Ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς όσους τονίσατε ότι χρειάζονται κανόνες για την καλύτερη κινητικότητα των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τις εταιρείε. Πράγματι αυτό θέλαμε. Θέλαμε να έχουμε αυτή την νομοθεσία διευκόλυνσης η οποία θα ε, παρέχει και ασφαλιστικές δικλείδες κατά της κατάχρησης, ασφαλιστικές δικλείδες που θα εγγυώνται το σεβασμό των δικαιωμάτων των μετόχων ε, και των εργαζομένων, που θα εγγυώνται ότι δεν ε, θα έχουμε φοροποφυγή, φοροδιαφυγή ή τη δημιουργία εταιριών προπετασμάτων, εταιριών γραμματοκιβωτίου. Ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκη αυτή η νομοθεσία, χρειάστηκε πολύ εμπειρογνωμοσύνη και όπως είπα και στην αρχή, χρειάστηκε και μεγάλη πολιτική βούληση. Επίσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ότι συνεργαστήκαμε σε ένα πνεύμα συμβιβασμού και βέβαια μας πίζει και ο χρόνος ε, στο τέλος. Είμαστε στο τέλος της θητείας μας, αλλά τα καταφέραμε. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη συνεργασία Πιστεύω ότι από κοινού παρουσιάζομαι μια καλή και ισορροπημένη πρόταση. Και ελπίζω ότι αύριο θα υπερψηφιστεί στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιώροβα. Η Ευελίν Ρέκνε τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε όποιος ε, έχει ασχοληθεί με το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο ε, πρέπει να είναι μαραθωνοδρόμος με ε, ικανότητες ταχείας με ικανότητες πρινταρίσματος όπως τα έλεγα. Γι' αυτό το λόγο εμείς ασχολούμαστε με το θέμα αυτό εδώ και πολλά χρόνια για να επιτύχουμε καλές προδιαγραφές στην Ευρώπη. Εμάς μας ενδιαφέρει ποιότητα και μέχρι και το τέλος, μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας αγωνιστήκαμε για να περάσει η δέσμη μέτρων. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Επίτροπο, ε, τους ε, διαπραγματευτές από τη Ρουμανική Προεδρία, την Καμπριέλα συγκεκριμένα, να ευχαριστήσω ε, τους ε, σκιώδης συγητές και κυρίως και τους συνεργάτες μας. Θα ήθελα αυτό το τελευταίο λεπτό να το εκμεταλλευτώ για να πω ότι ναι πράγματι έχουμε τώρα επιτύχει πάρα πολλά και σημαντικά αλλά το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η οδηγία πλαίσιο. Χρειαζόμαστε ένα οριζόντιο εργαλείο για τους εργαζόμενους έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειαζόμαστε και το περίφημο escalator έτσι ώστε να μπορεί να γίνει, να υπάρξει προσαρμογή ανάλογα με τις ε, καταστάσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε ε, και σας συζητήτρια και την Επίτροπο έκλεισε η συζήτηση αυτή και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Και συνεχίζουμε στην ημερήσια διάταξη και φτάνουμε τώρα στην ε, έκθεση του κύριου Στίσλαβ Κρασνοντεύσκη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή πρώτα. Παρακαλώ. Για τέσσερα λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου. Γιατί μετά από τρεις τριμερείς διαλόγους και ώρες διαπραγματεύσεων, καταφέραμε επιτέλους να καταλήξουμε σε μια μερική συμφωνία που θα ψηφιστεί αύριο. Δεν ήταν κάτι εύκολο. Εκφράστηκαν πολλοί φόβοι για το ταμείο αυτό. Φόβοι που εμένα μου φαίνεται ότι δεν έχουν καμία βάση. Αυτοί οι φόβοι, αυτές οι διαφωνίες, οι αντιδράσεις υπάρχουν ακόμα κάτι το οποίο μένα με εκπλήσει. Εγώ προσπάθησα να λάβω υπόψη μου τα επιχειρήματα όλων των πλευρών, όλων των συναδέρφων. του κύριου Μπούτικοφερ, για παράδειγμα, του κύριου Μαρτά, προσπάθησα να λάβω υπόψη μου τα επιχειρήματά τους και είχα την αίσθηση ότι οι συνάδελφοι αυτοί ήταν λίγο πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι θέτουν υπομφισβήτηση το κείμενο αυτό και βασίζονται ε, στα εξή δύο επιχειρήματα. Το ένα είναι ηθικής και το άλλο έχει να κάνει με τη φύση της κατεξοδότηση πράξης. Το ζήτημα ήταν, όσον αφορά την ηθική πτυχή, το μήπω, το Ταμείο αυτό αμφισβητεί τις σχέσεις μας με την Ατλαντική Συμμαχία, με το ΝΑΤΟ, που αποτελεί και την δομή που μα εγγυάται την ασφάλειά μας. Αυτό ερχόταν μάλλον από το αριστερό τμήμα του ημικυκλίου. Ακόμα και αν υπήρχαν ε, τέτοιες φωνές που ακούστηκαν και από το κέντρο και από τη δεξιά πτέρυγα του ημικυκλίου. Αυτά τα επιχειρήματα δεν έχουν βάση. Ο συμβασμός στον οποίο καταλήξαμε πιστεύω ότι αναγκάζει το Συμβούλιο να σέβεται απόλυτα τα όσα διαπραγματευτήκαμε. Είμαι επίσης πεπισμένος ότι η Επιτροπή, η Επίτροπος, είναι ικανοποιημένη και αυτή από τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε. Επιτρέψτε μου τώρα να παριθμίσω κάπως γρήγορα τι πέτυχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλο ότι το Ταμείο αυτό θα το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, ότι η τεχνολογία θα διακρίνεται ότι το επιπλέον ο κόστος δεν θα περιορίζεται, ότι θα υπάρχουν προϋποθέσεις προτιμησιακές στη συμμετοχή για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως και εκείνες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης και επίσης ότι θα υπάρχουν απαιτήσει ηθικής πάρα πολύ αυστηρές για οποιαδήποτε δράση χρηματοδοτείται από το Ταμείο αυτό. Συνεπώς, πετύχαμε πολλά από το Συμβούλιο. Αν συγκρίνουμε, δηλαδή, ότι προβλέπετε για το Ταμείο από το ΕΔΙΤΠ, αυτό που είναι, ας πούμε, για μένα πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να πετύχουμε ότι επιχειρήσεις που ελέγχονται από το κράτος αν υπάρχουν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλείονται από την χρηματοδότηση. Επίσης πετύχαμε ότι η αναφορά για στήριξη από το Ταμείο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Άμυνα για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί έτσι δείχνουμε ότι το Ταμείο δεν θέλει να στρατιωτικοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να προωθήσει τις εξαγωγές όπλων. Όχι, θέλουμε να στηρίξουμε την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα των εξοπλισμών. Και είμαι πεπισμένος ότι το Ταμείο αυτό θα επιτρέψει να δημιουργήσουμε νέα τεχνολογία και άμυνα υψηλού επίπεδου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που δεν καταφέραμε όμως να πετύχουμε από την άλλη μεριά εννοείται είναι μέσα στη φύση του Ταμείου, είναι η κατεξιοδότηση πράξη. Θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί το Ταμείο από την αρχή του 2021. Ίσως υπάρχουν και άλλα στοιχεία που θα έπρεπε να αναφέρει κανείς, αλλά εγώ αυτά ήθελα να πω μέχρι τώρα. Διατηρήσαμε τα πιο σημαντικά. Τα πιο σημαντικά επιχειρήματα αυτά της αριστεράς δεν στέκουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ευχαρι... Επόμενος ε, ομιλητής ε, εκ μέρους ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο πρόεδρος ο κ. Μακάλιστερ. Παρακαλώ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε, με το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο κάνουμε ένα μεγάλο βήμα έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα κοινά στοιχεία στην ε, έρευνα και στον, ε, στην αγορά ε, στρατιωτικών εξοπλισμών. Έτσι για να μπορούμε να οργανώσουμε την άμυνά μας. Ως εισηγητής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για το θέμα αυτό, ένα πράγμα κρίνω ιδιαίτερα σημαντικό. Το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο θέτει τα θεμέλια για καλύτερη συνεργασία και πάνω σε αυτό ε, μπορούμε να οικοδομήσουμε περαιτέρω σε θέματα ασφάλειας, ε, πολιτικής ασφάλειας, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση των ε, εθνικών ενόπλων δυνάμεων. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε καλύτερη στρατιωτική ικανότητα και σε τελική ανάλυση μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τους φόρους. Με το αμυντικό ταμείο βελτιώνουμε την αμυντική μας ικανότητα και εκ τούτου και την προστασία των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν καλώ όλους τους συναδέλφους αύριο το μεσημέρι να υπερψηφίσουν αυτόν τον κανονισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία, ε, κύριε Μακάλιστερ. Τώρα, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Πιανκόφσκα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, για άλλη μια φορά χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία ή που μας δίνετε ευκαιρία να συζητήσουμε για το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο. Δεν υπάρχει συνεργασία για τα θέματα αυτά στην Ευρώπη. Η πρόταση της Επιτροπής, από τότε που υπήρξε αυτή η πρόταση, είχαμε πολύ ουσιαστική δουλειά. Ε, σήμερα έχουμε μία ψηφωνία για την οποία ελπίζω ότι θα υπερψηφίσουμε αύριο τα βασικά στοιχεία του Ταμείου αποτελούν ορόσημο για την Μυντική Ένωση. Θα ήθελα ευθύ εξ αρχή να ευχαριστήσω την ε, διαπραγματευτική ομάδα της Ήτρε. Όλοι σας ε, είσαστε πολύ αφοσιωμένοι. Ο εισηγητής, η κυρία Γκροστέ, το κύριο Ρικέ, Μαρτάν Μπιουτικόφερ και βεβαίως ε, δεν πρέπει να ξεχνάω και τον κύριο Μακάλιστε. Σας ευχαριστώ όλους σας θερμά. Το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο θα ενισχύσει την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, θα βελτιώσει την αμυντική της ικανότητα και από την άλλη ε, θα βελτιωθεί η χρήση των ε, δημόσιων κοντιλίων. Με το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο χρησιμοποιούμε τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ευαισθητοποιήσουμε, να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα, αλλά και να επιφέρουμε καινοτομίες ε, βελτιώνοντας ε, την τεχνολογική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος κάνοντας την Ευρώπη μια πηγή ασφάλειας, ε, όχι ε, σε αντίφαση με τον ΝΑΤΟ, αλλά συμπληρώνοντάς του. Θα περιλαμβάνονται πάρα πολλά στοιχεία Γι' αυτά αγωνίστηκε σκληρά το Κοινοβούλιο. Θα αναφέρω λίγα εξ αυτών. Τα ανέφερε ο εισηγητή, αλλά θα τα πω και εγώ από την προοπτική τη Επιτροπή. Πρώτον, οι κανόνε Ευρωπαϊκή Ένωσης θα ισχύουν με βάση τον κανονισμό και την ενωσιακή ε, διακυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε με τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Ε, το ε, Κοινοβούλιο θα στηρίξει αυτό το Ταμείο. Δεύτερον, τεθεί το θέμα της ε, επιλεξιμότητας σε σχέση με το Ταμείο. Εδώ οι κανόνες είναι σαφείς. Μόνο οι ενωσιακές ε, εταιρείε, οι οποίες ε, σέβονται θέματα ασφάλειας στον εφοδιασμό και σε πολλούς άλλους τομείς, μόνο αυτοί θα μπορούν να συμμετέχουν. Δεν θέλουμε να εξαιρέσουμε κανένα, απλά ορίζουμε τις προϋποθέσεις για συμμετοχή για να διασφαλίσουμε ότι θα εξασφαλίζονται τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Αυτές οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι ευρωπαϊκές εταιρείε όταν ασχολούνται με έρευνα και ανάπτυξη σε τρίτες χώρες. Τρίτο θέμα, συνεργασία. Αυτό βρίσκεται στην καρδιά του Ταμείου. Εμείς δίνουμε κίνητρα με συγκεκριμένους κανόνες, προκαλώντας και την συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο δεν αφορά μόνο τους μεγάλους αμυντικούς ομίλους, αλλά και μικρούς παίκτες ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εμείς ελπίζουμε να ανοίξουμε την αλυσίδα την αμυντική. Τέταρτον, στο νομικό κείμενο καθίσατε σαφές ότι οι πράξεις θα πρέπει να είναι συμβατές ε, με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, όπως επίσης και με ηθικές αρχές που περιλαμβάνουν τα δίκαια αυτά. Το Κοινοβούλιο ζήτησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα ε, εκφραστεί επί των θεμάτων της ε, δεοντολογίας και επί των εμπειρογνωμόνων. Επίσης το Ταμείο αποκλεί δράσεις για την ανάπτυξη θανατηφόρων όπλων χωρίς ανθρώπινο έλεγχο. Εξάλλου, εμείς θα στηρίξουμε τις καινοτομίες το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα αυτό ε, βρίσκονται στην ίδια θέση, κυρίως όσον αφορά τις αποκαλούμενες disruptive τεχνολογίες. Αναφέρθηκε προηγουμένως από τον κύριο Σιγητή ότι ε, θα έχουμε τις ε, εφαρμοστικές πράξεις Έχουμε ένα κατάλογο που εισήχθη για να οριστεί το πλαίσιο του προγράμματος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη και πρόθυμη να έρχεται κάθε χρόνο στο Κοινοβούλιο για να συζητιέται το πρόγραμμα. Αυτή η προσέγγιση δεν αφορά μόνο θέματα άμυνας. Υπάρχουν και άλλα ε, προγράμματα και άλλες προτάσεις χρηματοδότησης που καταφεύγουν σε εφαρμοστικές πράξεις και που γίνονται δεκτά από το Κοινοβούλιο και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε Μπιενκόφσκα. Στην ε, συνέχεια, από την Επίτροπη Προϋπολογισμών ο κύριος Λαμασούρ. Για ένα λεπτό, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι εξ ονόματος Επιτροπής Προπολογισμών. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ όλους ε, όσους πέτυχαν αυτή την μερική συμφωνία και ιδίως την ομάδα του Κοινοβουλίου η κυρία Επίτροπος ανέφερε τα μέλη της για την Επιτροπή Προπολογισμών. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα από τα πιο ενωτόμα ε, έργα του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Αγωνιστήκαμε για πολλά χρόνια προκειμένου η άμυνα να μπορεί να αποφεληθεί από κονδύλια της Ένωσης και χαίρομαι ιδιαίτερα που η συμφωνία αυτή δίνει στο πρόγραμμα όλα τα μέσα για να πετύχει τη φιλοδοξία του και μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα μέσα του InvestEU και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αύριο θα το επιβεβαιώσει η Ολομέλη. Επίση χαίρομαι για το πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα που στέλνει αυτό το πρόγραμμα σε ένα τομέα που βρίσκεται στην καρδιά τη Εθνική Κυριαρχία. Αυτό το ταμείο μα δείχνει ότι η μεταφορά ορισμένων αρμοδιοτήτων στη Ένωση θα επιτρέπει να έχουμε περισσότερη ασφάλεια για να έχουμε και μικρότερο συνολικό κόστος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Λαμασούρ. Στη συνέχεια, εκ μέρου του ΕΛΚ, η κυρία Γκροστέτ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η τελευταία μου παρέμβαση στο κύκλο αυτό μετά από 20 ετή παρουσία και είμαι ικανοποιημένη που μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας απόψε γιατί ελπίζω ότι θα είναι ένα επιπλέον εργαλείο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω της ανάπτυξης της συνεργασίας. Πρόκειται για ιστορική στιγμή και αποφαλούμε να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κρασνοντεύσκη και την Επίτροπο, την κυρία Μπιένκοφσκα, που μας επέτρεψαν να πετύχουμε μια ταχεία συμφωνία. Ε, βέβαια, κάποιοι προσπάθησαν να κάποιοι να μπλοκάρουν ε, τις διαπραγματεύσεις για να έχουμε πραγματική βιομηχανική πολιτική στον τομέα της άμενος και κάτι που κανείς δεν φανταζόταν δυνατό το πετύχαμε. Έτσι λοιπόν, ε, έχουμε μια πολύ καλή συμφωνία που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις και στο επόμενο κοινοβούλιο θα πρέπει να ψηφίσει τον προπολογισμό των 13 δισεκατομμυρίων την περίοδο 2021-2027. Θα πρέπει να προσελκύσουμε τα καλύτερα προγράμματα και τα πιο καινοτόμα από την πλευρά των κρατών μελών και τη βιομηχανία. Αυτό το Ταμείο απαντά στις ανησυχίες των πολιτών μας για την ηθική, για την απαγόρευση των θανατηφόρων οπλικών συστημάτων. να Έχουμε επιχειρήματα απέναντι σε κάποιε ειρηνικέ ε, ιδεολογίε που ε, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Αυτό το Ταμείο θα επιτρέψει στην Ευρώπη να ενισχύσει την αυτονομία τη σε στρατηγικό και τεχνολογικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μία ανεξάρτητη ικανότητα με χρηματοδότηση προ τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Αυτή η αρχή τη στρατηγική αυτονομία, είναι ζωτική σε πολλού άλλου τομεί. Στο διάστημα στην υγεία, την ενέργεια, τα τρόφιμα και βεβαίω στην ασφάλεια και στην άμυνα. Γιατί σε έναν όλο και πιο ασταθή κόσμο θα πρέπει να βασιζόμαστε στην ένωση με τι δικέ μας δυνάμει. Έτσι θα έχουμε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση που θα επιτρέψει να προστατεύσει καλύτερα την ασφάλεια των κρατών μας στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κροστέτ, και σας ευχόμαστε ότι καλύτερο στο μέλλον. Είπατε μετά από 25 χρόνια είναι η τελευταία σας παρέμβαση αυτή. Ωραία. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Εντουάρ Μαρτά, παρακαλώ. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως και καταλαβαίνω ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο κατάφεραν να φτάσουν σε αυτήν την συμφωνία και χαίρονται, αυτό θέλανε και δεν υπάρχει κατεξουσιοδότηση πράξη. Κάτι που μπορεί να φαίνεται ένα τεχνικό στοιχείο για πολλού, αλλά όχι, γιατί είναι θέμα ελέγχου από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άρα των πολιτών για ένα πρόγραμμα 13 δισεκατομμυρίων και για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Φυσικά και στηρίζω τις τροπολογίες που θα ψηφίσουμε αύριο και ιδιαίτερα το άρθρο για την απαγόρευση κάποιων όπλων, το άρθρο 11 επίσης, γιατί πράγματι δεν είναι δυνατόν απλώς να αναφερόμαστε στο διεθνές δίκαιο, γιατί υπάρχει εμφυσιμία εδώ. Για παράδειγμα, ο λευκός φόσφορος, η χρήση του για πυρομαχικά επιτρέπεται. Αν όμως χρησιμοποιηθεί χωρίς ε, διακρίσεις εμπριστικά, αυτό το καταδικάζει η ίδια σύμβαση της Γενέβης. Και έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις που έχει καταδικάσει ΙΕ ε, στην Γάζα, για παράδειγμα. Έπειτα, το απεμπλουτισμένο ουράνιο και εδώ, σαν όπλο απαγορεύεται στο Βέλγιο. Δεν ρυθμίζεται όμως αλλού και ούτε αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο. Εφόσον λοιπόν ό,τι δεν απαγορεύεται επιτρέπεται, θα έπρεπε να έχουμε ένα κατάλογο με συγκεκριμένον εξοπλισμό για τον οποίο δεν πρέπει να επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, για τις εξαγωγές όπλων. Δεν είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κυρώνει την προσέγγιση που θέλει το Συμβούλιο να είναι όλα στην διακριτική ευχαίρεια των χωρών μελών. Είναι θέμα ερμηνείας. Πού είναι τα 8 κριτήρια του 2008 και η συμφωνία για την εμπορία των όπλων που έχουν επικυρώσει όλε οι χώρε. Αυτά μπορεί εσά να σα φαίνονται λεπτομέρειε, για μένα έχουν τεράστια σημασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρτά. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ντομινίκ Ρικέ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον εισηγητή μας, τον κύριο Κρασνοντέψκι, για την υπομονή του και για τη δουλειά του. Επανέρχομαι στην ηθική αυτή τη πρόταση, τα ανέφεραν και η Επίτροπο και ο εισηγητή, αλλά πολιτικά θέλω να πω ότι πρόκειται για μια τεράστια πρόοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιστορία θα το θυμάται αυτό. Από το 54, το 1954 προσπαθούμε και όμως δεν καταφέραμε να έχουμε την κοινότητα άμυνας και τώρα το 2019 επανερχόμαστε και προσπαθούμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις αυτής της κοινότητας που απέτυχε. Τώρα λοιπόν όλα αυτά τι δείχνουν. Δείχνουν εμπιστοσύνη, δείχνουν αλληλεγγύη. Να μην υπάρχει επικάλυψη σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης στην άμυνα, μείωση του κόστους, η οικονομία κλίμακος. Το γεγονός ότι ζούμε σε έναν κόσμο όλο και περισσότερο αβέβαιο, με μεγάλη αστάθεια, καλό είναι να μπορούμε να διασφαλίζουμε την προστασία μας σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το Ταμείο αυτό θα μας επιτρέψει καλύτερη ενσωμάτωση των εργαλείων των αμυντικών θα μας βοηθήσει να κάνουμε οικονομίες και θα υπάρξει και μία παρετέρω ολοκλήρωση. Κρίμα που υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες σαν στόχο έχουν να εμποδίσουν τη συμφωνία σε τριμερή διάλογο. Κι όμως είχαμε καταφέρει να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία και μας εκπλήσει που ένα τόσο σημαντικό θέμα τελικά το χειριζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Εμεί θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς που πιστεύουν στην Ευρώπη σε μια περισσότερο δυνατή Ευρώπη. Α φροντίσουμε να έχουμε μια πιο δυνατή Ευρώπη που να προστατεύει ακόμα καλύτερα τους πολίτες της. Να έχουμε αυτό το αμυντικό ταμείο ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και την δικιά μας την κυριαρχία, την βιομηχανική και την αμυντική και συγχρόνως να διασφαλίσουμε και την προστασία των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Ρικέ. Στη συνέχεια, εκ μέρου της ΓΚΟΕ, έχουμε την Μαρίσα Ματίας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο ζήτημα και μπορείτε να μιλάτε για χρηματοδότηση, αλλά να δώσουμε 13 δισεκατομμύρια από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα σημαίνει ότι αφαιρούμε 13 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα σημαίνει ότι θα ανταλλάξουμε την ελληνική τη συνοχή, τα μέτρα που προστατεύουν την ποιότητα ζωή των Ευρωπαϊκών πολιτών για να επενδύσουμε σε πιο αποτελεσματικά οπλικά συστήματα. Οι τεχνικές λύσεις ε, δεν αποτελούν ε, παρά ε, ουσιαστικά μια πρόφαση για την πώληση όπλων. Χρειάζονται ασφαλή Ευρωπαίοι, όμως στην απασχόληση, στις δημόσιες υπηρεσίες, σε ένα βιώσιμο μέλλον. Τίποτα δεν εμποδίζει τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν στον τομέα της άμυνας. Με τον ίδιο τρόπο, τίποτα δεν αιτιολογεί να δημιουργηθεί ε, μια νέα γραμμή του προπολογισμού ε, που ούτε καν σέβεται τα όσα εγγράφονται στη συνθήκη. Είναι μια πολύ ακριβή επιλογή και πολύ πιο ακριβή από τα 13 δισεκατομμύρια που έχουν εγγραφεί εδώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ματίας. Στη συνέχεια για τους πράσινους, ο κύριος Μπουτικόφερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι, το γεγονός ότι στην Ευρώπη πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την κοινή ασφάλεια. Αυτό είναι το σημείο κίνησης της επιχειρηματολογίας μου. Γι' αυτό λοιπόν ένα αμυντικό ταμείο το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παίξει ε, θετικό ρόλο. Όμως σε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις δεν πετύχαμε το εφικτό. Η επικάλυψη, η ανεπάρκεια θα εξακολουθούν να υπάρχουν στην ε, αγορά των εξοπλισμών το γεγονός ότι σπαταλήσαμε την ευκαιρία που μας προσφέρθηκε. Αυτό ε, δεν οφείλεται στον εισηγητή ε, που θέλω να τον επενέσω γιατί πραγματικά ε, είναι πνεύμα αντιλογίας, πρέπει να το πω αυτό και μερικές φορές μου κάνει και κέφι το να διαπληκτίζουμε μαζί του για το θέμα της πραγματικότητας και του ΝΑΤΟ. Τέλος πάντων, από τον ε, κύριο Ρουκέ και από την κυρία Γκροστέτ ε, άκουσα ξεκάθαρα του ΣΥΔΑ να εκπροσωπούν την, ε, τα γαλλικά λόμπι εξοπλισμών και την ε, στρατιωτικοποίηση, της σχετική ιδεολογία. Αυτό λοιπόν που έχουμε τώρα είναι ένα αμυντικό ταμείο ε, του οποίου η δεοντολογία και οι αρχές περιοντολογίες είναι απλά μία βιτρίνα. Ένα αμυντικό ταμείο που πολύ σωστά είπε ο κύριος Μαρτά, ένα ταμείο σε 7 χρόνια θα διαθέσει 13 δις ένα αμυντικό ταμείο που θα οδηγήσει τελικά ε, στο να έχουμε περισσότερες εξαγωγές εξοπλισμών. Ένας τέτοιος ευνουχισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι όνειδος. Αλλά παρόλα αυτά σημειώθηκε μια καλή ουσιαστική επιτυχία ότι δεν θα δοθούν χρήματα για τους, ε, για τα ρομπότ δολοφόνους. Δεν αρκεί όμως αυτό. Και γι' αυτό εμείς ε, θα καταψηφίσουμε. Κατά τα άλλα, να σας προειδοποιήσω για άλλη μια φορά όσον αφορά την ιδεολογία της ε, στρατηγικής αυτονομίας. Όποιος προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να παρουσιάσει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, είναι απλά εθεροβάμων. Ευχαριστώ κύριε Μπουτικόφερ. Στη συνέχεια, ο κύριος Μπουλόκ για δύο λεπτά έχετε το λόγο. Πρόεδρε, προκειμένου να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, η Επιτροπή Γιούνκερ θέλει να χρηματοδοτήσει έργα άμυνος που θα κοστίζουν 13 δισεκατομμύρια ευρώ τεχνολογία για τετρών, επικοινωνίες με δορυφόρους, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, εποπτεία στη θάλασσα. Συνεχίζει να εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση προς μια ολοκληρωτική ένωση και τελικά προς μια στρατιωτική. Η Κομισιόν προσπαθεί να παρουσιάσει αυτή την εξέλιξη που μια ειρηνευτική διαδικασία. Όμω είναι σαφόφωνα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υποστηρικτέ τη έχουν έναν στρατό κατά νου. Ο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν ε, ενθάρρυνε τη δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Στρατού πρόσφατα για την υπεράσπιση τη Ευρώπη. Πώ μπορεί κάποιο να δημιουργήσει ένα μοσπονδιακό στρατιωτικό ε, έργο που θα συμμετέχουν 27 ε, κράτη και 24 γλώσσε, ε, όπω συνήθισε να λέει η Μάργαρετ Θάτσερ, δεν έχει χρήματα παρά τα χρήματα που κερδίζουν οι ίδιοι άνθρωποι. Κάποια στιγμή που, τη στιγμή που είναι σε κρίση το ευρώ και γίνονται περικοπές για την ανάπτυξη, ε, τώρα, η έλλειψη ανταγωνιστικότητα τη ε, βιομηχανία ανησυχεί του πολίτε, όπως και αν άνθρακα. ένα πανευρωπαϊκό στρατός ε, θα είναι η τελευταία ευρωπαϊκή καταστροφή σε αντίθεση με τη Ρωσία ή τη ΕΙΠΑ. Δεν είναι ένας νέο παράγοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε και την ψηφοφορία για το Brexit ε, και ε, την ε, κυβέρνηση της Ιταλίας που θα αποθαρρύνουν την περαιτέρω ομοσπονδιοποίηση. Εδώ έχουμε ένα σύνολο γραφειοκρατών που λαμβάνουν αποφάσεις για την άμυνα, για τον πόλεμο και την ειρήνη. Εμείς είμαστε κατά της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού στρατού και ελπίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θα συνειδητοποιήσουν ότι να δίνουν περισσότερες αρμοδιότητες στην Κομισιόν είναι λάθος και είναι η τελευταία μου ομιλία σε αυτό το κοινοβούλιο και ε, απευθύνω έκκληση να απομακρυνθείτε από ένα ευρωπαϊκό υπερκράτος και δεν θα υπάρξει κανένα καλό από τη δημιουργία στρατού και ελπίζω ότι οι εκλογές για το νέο κοινοβούλιο θα ανατρέψουν αυτή την τάση και θα προωθήσουν το σεβασμό του έθνους κράτους και της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπουλόκ. Και Καλή επιτυχία για το μέλλον. Να σας ευχηθώ. Στη συνέχεια περνάμε στον κύριο Μπούζεκ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλουμε να ενισχύσουμε τον αμυντικό πυλώνα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Και πρέπει να θυμηθούμε ότι η βιομηχανία άμυνας δεν είναι μόνο η ασφάλεια, αλλά είναι και η ανάπτυξη της βιομηχανίας γενικότερα στην Ευρώπη. Ως πρόεδρος της Αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής είμαι ικανοποιημένο όχι μόνο λοιπόν για την ανάπτυξη της άμυνας, αλλά και της βιομηχανίας άμυνας. Περί τίνος πρόκειται. Πρώτα απ' όλα πρόκειται για την συμμετοχή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Δεύτερον, πρόκειται για την ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης και πρόκειται και για ενθάρρυνση των χωρών μελών να συνεργαστούν μεταξύ τους σε σχέση με τις παραγγελίες και τις προσφορές. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό επιχείρημα στην δικιά μου την περιφέρεια. Έτσι θα μπορέσουμε, πιστεύω, σύντομα να κάνουμε τους Ευρωπαίους να υποφεληθούν από τεχνολογικές λύσεις οι οποίες θα έχουν δημιουργηθεί από τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις της δικιάς μου περιφέρειας. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή μας, τον κύριο Κρασνοντεύσκη, ο οποίος πάρα πολύ καλά βοήθησε στις διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και όλους τους συνεισηγητές, όπως επίσης και την κυρία Γκροστέτ, η οποία ήταν προηγουμένως η συγγήτρια της δικιάς μας έκθεσης για το ίδιο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάνουμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πουσέκ, ο επόμενος, ο Βίκτορ Μποστινάρου. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κυρία, κυρία Επίτροπε, να ξεκινήσω από εσά. Σα ευχαριστώ κύριε Σιγητά για τον εξαιρετικό τρόπο που διαπραγματευτήκατε σε ένα κόσμο που έχουμε αστάθεια και πολλές ευρυδικές και νέες απειλές. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παγιώσει το ρόλο της ως παγκόσμιο παίκτη που θα ασκεί επιρροή. Σήμερα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την άμυνα αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για όλους τους πολίτες μας και ε, ε, γι' αυτό βρήκε απήχηση. Η ανάπτυξη της ε, κοινή πολιτικής άμυνας είναι μία από τις κύριες συνεισφορές στην εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σκόπος της νομοθετικής πρότασης που έτυχε διαπραγμάτευσης με το Συμβουλίο είναι να ιδρυθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, έτσι ώστε να απαντήσει στις αυξανόμενες προτεραιότητες της άμυνας και της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να να αρχίσουμε να ε, απαντάμε στον κατακαιρματισμό του τομέα της άμυνας ε, και να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, ε, να ενθαρρύνουμε την ε, συνεργασία και την κοινή απόκτηση εξοπλισμών. Επίσης, όπως ανακοινώθηκε, είχαμε κύριες προτεραιότητες κλειδί της δικής μου πολιτικής ομάδας για το τομείο αυτό. Εμείς αγωνιζόμαστε για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αμυντική βιομηχανία και στην πρόθεση μιας ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς ε, για ε, τα μέσα άμυνας. Αγαπητοί συνάδελφοι, και πάλι να υπογραμμίσω την ανάγκη να συνεχίσουμε τη διαδικασία της ε, προώθησης μιας παγκόσμιας τάξης βάσει κανόνων, έτσι όπως αναφέρεται στην Χάρτα 1 και να παγιώσουμε τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, καθώς αυτό αποτελεί τη μόνη εγγύηση ασφάλειας στην Ήπειρό Είχα την ε, το προνόμιο να εργαστώ στο φάκελο αυτό τα τελευταία χρόνια και θα ήθελα να σας συστήσω να υπερψηφίσετε αύριο. Και καθώς αυτή είναι η τελευταία μου ομιλία στο κοινοβόλιο, επιτρέψτε μου να πω σε όλους σας ευχαριστώ καρδίας για αυτά τα 12 χρόνια τα οποία εργαστήκαμε για το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα. Κυρία Γκροστέτ, ας ε, παραμείνουμε ειρηνικοί αλλά ποτέ αγαθοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μποστινάρου. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Φερέιρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, 13 δισεκατομμύρια ευρώ τόσα ε, θέλει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα των ε, μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων σε 7 χρόνια. Αυτά αφαιρούνται από τις επενδύσεις στην καταπολέμηση στόχη την πρόθεση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Είναι πόροι που θα προωθήσουν τώρα τον πόλεμο, θα χρηματοδοτήσουν την εξοπλιστική βιομηχανία, τροφοδοτώντα μια κούρσα στρατιωτικοποίησης. Ε, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ανοίγεται και την πότρη του προγράμματος έρευνας ε, για, όχι αποκλειστικά για ειρηνικού ε, και μη στρατιωτικού σκοπούς και θα χρησιμοποιήσετε τα δίκτυα μεταφορών για τη στρατιωτική κινητικότητα. Όποιο προωθεί τον πόλεμο και τροφοδοτεί αυτή τη βιομηχανία δεν μπορεί να πετύχει την ειρήνη. Έτσι λοιπόν αυτή η νομοθεσία δεν σέβεται ε, τους λαούς. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο συνεργασίας που να έγκυται στις ε, αξίες της ειρήνης. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Φεραίρα. Και τώρα ο κύριος Μπουτικόφερ έχει θέσει μια μπλε κάρτα. Δέχεστε παρακαλώ. Κύριε Φερέιρα, υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας. Σας μιλώ φιλανδικά. Δέχεστε την μπλε κάρτα από τον κύριο Μπουτικόφερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φερέιρα, το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι στραφήκατε κατά της ε, στρατιωτικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πώς μπορείτε να μας εξηγήσετε ότι η δική σας η πολιτική ομάδα, η ΓΚΟΕ, σε όλες αυτές ε, τις διαπραγματεύσεις των πολλών μηνών δεν εμφανίστηκε ούτε μία φορά ένας έστω ε, ευρωβουλευτής για να συζητήσει. Και δεν καταλαβαίνω πώς τολμάτε να στρέφεστε κατά του μιλιταρισμού και δεν έχετε κάνει τα μαθήματά σας. Κύριε Μπουτικόφερα, αύριο θα επιβεβαιώσετε ότι δεν θα είναι με την υποστήριξη αυτή τη ομάδα που αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα που θέλει να διθέσει 13 δισεκατομμύρια ευρώ ε, στην εξοπλιστική μηχανία θα εγκριθεί. σω ε, με κάποιε ψήφου από τη δική σα πλευρά, δεν ξέρω, θα δούμε. Σίγουρα με τι ψήφου τη Σοσιαλδημοκρατία και όλη δεξιά. Και φυσικά δεν αγνοώ τη σύνθεση αυτού του οίκου, όπω και εσεί. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι θέσει μα είναι μη ψηφικέ ακόμη. Και λέω ακόμη γιατί νωρίτερα ή αργότερα γρήγορα και μάλλον νωρίτερα θα είναι πλειοψηφικέ ε, απόψει ε, και εμεί θα ανατρέψουμε αυτή την κούρσα εξοπλισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι εσεί κάπω έχετε ανεχθεί στο παρελθόν αυτέ τι ε, στρατιωτικέ περιπέτειε. Ja sitten edustaja Inrik Taransa puheenvuoro, niin hänellä on minuutti. Olkaa hyvä, edustaja Taran. Ο κύριος Ταράν, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον ε, συνάδελφό μου, κύριο Μπίτι Κόφα. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι παρότι άσκησε κριτική κατά αυτής της πρότασης και σωστά έπραξε, φαντάζομαι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι το Ευρωπαϊκό Αμαντικό Ταμείο έρχεται ε, πολύ καθυστερημένα και είναι και πολύ λίγο γιατί δεν κατορθώσαμε να νομοθετήσουμε για να υπάρχει μια, ε, ε, ένας ευρωπαϊκός στρατός που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να υπερασπιστεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα άλλα, υποστηρίζω την έκθεση όσον αφορά την αίρεσιμότητα, ότι δηλαδή πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα. Ε, προς τον κύριο Μπούλοκ ε, θα ήθελα να πω ότι η ο Ευρωπαϊκός Αμυντικός Στρατός ε, θα υπάρξει, θα μιλάει αγγλικά. Δυστυχώς ε, λόγω αυτής της περιπέτειας του Brexit δεν θα υπάρξει Βρετανός διοικητής, αλλά θα υπάρξει αυτός ο στρατός. Και προς τον κύριο Φαρέρη, θέλω να πω ότι τα τρία δις είναι τίποτα, ψίχουλα. Ακόμα και ο προπολογισμό ε, της ε, Λετωνία είναι πολύ μεγαλύτερο. Ο κύριος Καστάλντο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ψηφοφορία αύριο για το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο έρχεται στο τέλο μια μακρά και περίπλοκη διαδικασία και ευχαριστώ τον εισηγητή. Ε, δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά που μα οδήγησαν μέχρι εδώ. Εγώ ήμουν και ο εισηγητής, αλλά θέλω να ζητήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει να ελέγχει ε, την ε, εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου. Αύριο δεν είναι το τέλο, αλλά είναι η αρχή μια ε, νέα αμυντική πολιτική. Το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να είναι παίκτη και όχι παρατηρητής. Εγώ ήμουν υπέρ και γενικά η δική μας η ομάδα ήταν υπέρ των ε, κατεξοδότηση πράξεων. Ορισμένες τροπολογίες ε, πέρασαν το, στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να υψώνει τη φωνή του για να υπάρχει ένα ε, όραμα πραγματικά ευρωπαϊκό που θα επιτρέπει τρία στάδια με πνεύμα του ανταγωνισμού θα πρέπει να βελτιώσουμε τις ε, τεχνολογίες μας. Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να μην υπάρχουν ε, άμεσες απευθείας αναθέσεις. Ε, εμείς έχουμε εκφράσει επιφυλάξεις για κάποια κριτήρια, αλλά θέλουμε να ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα εφαρμοστούν χωρίς τιμωρητική διάθεση. Θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι εμείς δεν θέλουμε να έχουμε ένα εργαλείο το οποίο με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρηματοδοτεί λάθους στόχους. Δεν θέλουμε να υπάρχει συνεργασία με άλλους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά την παραγωγή και την έρευνα. Δεν θέλουμε ε, να διαταράσσεται η αλυσίδα παραγωγής ε, με το να αποκλείονται κάποιες χώρες. Ε, επίσης δεν θέλουμε σε τελική ανάλυση αυτό το ταμείο να ε, χρηματοδοτεί θανατηφόρα όπλα χωρίς ελεγχό η πρόεδρος διακόπτη. Ο κύριος Καστάντο μιλάει με ένα ρυθμό απίστευτα γρήγορο. Πάση περιπτώσει, θέλουμε λοιπόν να ανοίξουμε την πόρτα για έναν ευρωπαϊκό στρατό, ακόμα και εάν ε, ε, αναφέρονται οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου στις συνθήκες. Εμείς ε, θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε αυτό το ταμείο, ένα ταμείο το οποίο θα διευκολύνει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα διευκολύνει την άμυνα και την ε, ασφάλεια, ένα ταμείο το οποίο δεν θα στρέφεται κατά άλλων, αλλά ούτε θα θέλει να προστατεύει ιδιαίτερα κάποιους, ένα ταμείο το οποίο θα είναι ανοιχτό για άλλες συνέργειες. Τέλος, το ταμείο αυτό θα πρέπει να βοηθήσει να ξεπεραστούν τα κενά, χωρίς να ξεχνάμε ότι οι τελικοί χρήστες ε, θα είναι οι δικοί μας οι άντρες ε, και οι γυναίκες ε, και όλοι εκείνοι που βρίσκονται και σε καθεστώς πολέμου. Πρόεδρος, κοιτάξτε, οι διερμηνείς πραγματικά τώρα εξεπέρασαν τον εαυτό τους, γιατί δεν υπάρχει και όριο στην ταχύτητα. Μιλάτε τόσο πολύ γρήγορα. Αν έχετε την καλοσύνη, λίγο πιο, πιο αργό ρυθμό, λέει η πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Γκάλερ. Παρακαλώ κύριε Γκάλερ. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια σημαντική συνεισφορά έτσι ώστε οι πολίτες μας να προστατεύονται από εξωτερικές απειλές. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει αυτό το ταμείο ε, για να μπορεί να αξιολογηθεί η ασφάλεια και να γίνουν περισσότερα πράγματα. Το βρίσκω πάρα πολύ λυπηρό το ότι κάποιοι από αριστερά αλλά και μέχρι δεξιά ε, δεν θέλουν να προσφέρουν αυτή την καλύτερη προστασία στους πολίτες μας. Αυτό είναι ολιγορία. Ολιγορία κατά των πολιτών μας που τους αξίζει καλύτερη άμυνα ολιγορία και έναντι των στρατιωτών μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή παραδείγματος χάρη στο Μαλί, ε, στη Σομαλία, στη Μεσόγειο υπερασπίζονται τα συμφέροντά μας. Έχουν το δικαίωμα να έχουν τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίζουν υγιείς στις πατρίδες τους. Τέλος, αναφέρομαι στο Συμβούλιο και στα μεμονωμένα κράτη-μέλη και στην Επιτροπή. Στο μέλλον εσείς θα κληθείτε να αποδείξετε ελέγξετε ότι τα 13 δις που προβλέπονται για τον αμυντικό αυτό προπολογισμό θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από κοινού για αγορές, ε, για εξοπλισμούς, ε, για βελτίωση της ικανότητας. Τώρα πρέπει να αποδείξετε ότι ε, τα 210 δις ευρώ στο μέλλον θα χρησιμοποιούνται καλύτερα οι πρωτεύουσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν και όχι να θέλουν να καταφύγουν σε προγράμματα όπως το ΕΦΚΑΣ ή τα τεθωρακισμένα μάχης. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να εξηγήσετε στους πολίτες μας τελικά τι εξυπηρετούν όλα αυτά. Από το σύνθημα στρατηγική αυτονομία θα πρέπει να περάσετε σε μια συνεπή αμυντική πολιτική, πολιτική εξοπλισμών, έτσι ώστε οι πολίτες μας και η βιομηχανία μας να κατανοούν περί πρόκειται. Ε, το ταμείο για το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο είναι το, μόνο το πρώτο βήμα και κατά τα άλλα θα χαιρόμουν πάρα πολύ ε, το πώς θα, να δω πώς θα ψηφίσω ο κύριος Μπούλμαν από τον ε, πρόεδρο μια τόσο μεγάλη πολιτική ομάδα σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, μπορεί κανεί να περιμένει και μια προσωπική τοποθέτηση. Ο κύριος Ροζάτης στη συνέχεια για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. κύριε Επίτροπε, σήμερα συζητάμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την ασφάλεια της Ευρώπης, ε, μια αγορά δημόσιων κονδυλίων ε, για την απόκτηση αμυντικών μέσων. Αυτό είναι κατακαιρματισμένο ε, στην Ευρώπη. Μόλις το 16% αυτών των ε, δημόσιων διαγωνισμών υλοποιούνται από δύο ή περισσότερα κρατημέλη. Το αποτέλεσμα είναι ότι το επίπεδο συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στο απαιτούμενο επίπεδο. και φυσικά ε, η ασφάλεια αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας και υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις ε, όπως η επιθετική πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ο μουσουλμανικός ε, εξτρεμισμός και απαιτούν να ενισχύσουμε τις αμυντικές ικανότητες της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ακριβώς αποτελεί ένα μέσο το οποίο θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Σε αυτό το πλαίσιο η συνεργασία στο βιομηχανικό τομέα είναι πάρα πολύ σημαντική και θα μας επιτρέψει την ανάπτυξη του κλάδου στα κράτη-μέλη. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαθέτει 13 δισεκατομμυρία ευρώ. Ένα ποσό που θα επιτρέψει την ενίσχυση των ικανοτήτων ε, στην έρευνα και στην κοινοτομία στον αμυντικό κλάδο. Θα πρέπει να διατηρήσουμε μια ισορροπία στην κατανομή των κορτιλίων ε, για να μπορέσουμε ε, να προωθήσουμε το δυναμικό όλων των χωρών και αναφέρομαι και στις μεγάλες χώρες αλλά και στη χώρα μου στην Πολωνία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρωσάτη. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Κατσδιάη. Τρεις έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Πόσπεσιλ πρώτα απ' όλα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσωπικά όλη τη συζήτηση και θα την στηρίξω. Πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη. Αυτές οι επενδύσεις θα ενισχύσουν την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης θα ενισχύσουν την αμυντική βιομηχανία. Θα είναι κάτι πολύ σημαντικό γενικότερα για την οικονομία. Τέτοια προγράμματα δεν είναι δυνατόν βέβαια να απειλούν τη συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αποτελούν μια εναλλακτική λύση διαφορετική από το ΝΑΤΟ. Εμείς στην Τσεχία πιστεύουμε ότι η συνεργασία με το ΝΑΤΟ είναι ζωτική σημασίας. Οπότε πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση, αλλά η συνεργασία με τον ΝΑΤΟ να ξέρουμε ότι είναι το πιο σημαντικό. Πρώτος, ευχαριστούμε κύριε Πόσπισιλ. Ο κύριος Μαριάς τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. 13 δισεκατομμύρια ευρώ στο ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας. αυτό σημαίνει λιγότερα χρήματα στον προϋπολογισμό της ευρωπαϊκής ένωσης για την υγεία την παιδεία τις υποδομές την εκπαίδευση την κατάρτιση την αντιμετώπιση της φτώχειας. θεωρώ ότι αυτό το ποσό επί της ουσίας θα μπει στην υπηρεσία των μεγάλων πολεμικών βιομηχανιών της ευρωπαϊκής ένωσης που ως γνωστόν πουλάνε όπλα ακόμη και στην τουρκία ακόμη και στη σαουδική αραβία. στην πράξη τι γίνεται; ζήτησε ο τραμπ να βάλει η ευρωπαϊκή ένωση το χέρι στην τσέπη για τα θέματα της άμυνας. αυτό είναι όλο το θέμα. και πλέον ερχόμαστε να υπηρετήσουμε αυτή την πολιτική μετατρέποντας σε όλο και πιο στρατιωτικοποιημένη την ίδια την ευρωπαϊκή ένωση. και γι' αυτό αυτό που θα συμβεί στην πράξη είναι να γίνονται όλο και πιο πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις από πλευράς ευρωπαϊκής ένωσης στον τρίτο κόσμο. θεωρώ ότι τα κονδύλια αυτά πρέπει να πάνε κυρίως για τη στήριξη της ίδιας της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ευχαριστούμε κύριε Μαριά. Παρακαλώ. Κύριε Σόσνιερτς. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε αυτά που είπε ο καθηγητής Κρασνοντεύσκη, ότι πρόκειται για ένα παραπάνω βήμα για μια Ευρωπαϊκή Ένωση της Άμυνας. Και αρκεί να ακούσουμε την κυρία Κροστέτ για να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μια σε βάθος ολοκλήρωση. Καταλαβαίνω ότι οι Γερμανοί προσπαθούν να πετύχουν περισσότερα. Χάσαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οπότε τώρα βρίσκονται στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και δρούν ανάλογα. Πώς όμως θα υποφεληθεί η Πολωνία. Ουσιαστικά καταστρέφουμε την ανεξαρτησία μας. Χάνουμε τον έλεγχο του δικού μας στρατού. Η έρευνα και ανάπτυξη που μπαίνουν σε κοινό πλαίσιο σημαίνει ότι χάνουμε τον έλεγχο της δικιάς μας έρευνας και ανάπτυξης τι θα γίνει στις χώρες οι οποίες τελικά δεν θα έχουν το δικό τους στρατό. Φτιάχνουμε ένα τέταρτο Ράιχ της Γερμανίας. Πρόεδρος, τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, για τα σχόλιά σας, για τις παρατηρήσεις σας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με τίποτα δεν ήταν εύκολη η υπόθεση αυτή, δεν ήταν εύκολο να συμφωνήσουμε μεταξύ μας τα τρία ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι όλους που με τόση αφοσίωση προσπαθήσετε να ε, καταλήξουμε σε μια καλή λύση. Σε δύο πτυχές θα αναφερθώ μόνο. Πρώτον, για τη συνεργασία γιατί πολλοί από εσά αναφέρθηκαν στο ποσό, στα χρήματα. Θέλω να σας πω και πάλι ότι η έλλειψη συνεργασίας στον τομέα της άμυνας κοστίζει και το κόστος αυτό είναι ανάμεσα στα 25 με τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο επειδή δεν υπάρχει συνεργασία στον αμυντικό βιομηχανικό τομέα. Έπειτα, για την εξαγωγή όπλων, επειδή Κάποιοι από εσά το έθεσαν. Και εδώ είναι σαφές το θέμα. Έχουμε συζητήσει πολύ γι' αυτό. Είναι καθαρά αρμοδιότητα των χωρών μελών. Δεν αλλάζει αυτό με τίποτα με τον κανονισμό. Δεν αυξάνουμε την εξαγωγή όπλων. Αυτό που θέλουμε και αυτή που είναι η πρόθεσή μας είναι να μειωθεί η εξάρτησή μας από τρίτες χώρες. Η τεχνολογία μας να μην εξαρτάται από τρίτες χώρες. Η συνεργασία θα βοηθήσει σε αυτό. Η μείωση της τεχνολογικής μας εξάρτησης είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία του φακέλου αυτού. Και είμαι σίγουρη ότι η άμυνα θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μιλάμε ακόμα για την ε, αμυντική βιομηχανική συνεργασία. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαίρεται για την συμφωνία ε, στην οποία καταλήξαμε μετά τους τριμερείς διαλόγους. Και ελπίζω αύριο να υπερψηφιστεί η πρόταση αυτή. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ όλους, τον εισηγητή, τους όδες εισηγητές, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ίτρε, τον κύριο Μπούτσεκ, γιατί είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σκληρή δουλειά. Δεν ήταν εύκολο, αλλά νομίζω ότι η συμφωνία είναι ικανοποιητική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Επίτροπο ε, και τώρα λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο και πάλι στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης η οποία κατέδειξε ότι δεν ε, συμβίπτουν οι απόψεις μας. Στους σοσιαλδημοκράτες ε, εκφράστηκαν από πλευρά τους διαφορετικές απόψεις ε, και στο επίπεδο των, στο μέτωπο των πρασίνων και εκεί διαφορετικές απόψεις. Ε, υπάρχουν και διαφορές ανάμεσα στα κράτη. Υπάρχουν κράτη όπου δεν υπήρξαν εισβολές ούτε κατοχή εδαφών. Από την άλλη όμως υπάρχουν κράτη όπως οι χώρες της Βαλτικής και χώρες ε, της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που εξακολουθούν να αισθάνονται υπό απειλή. Ναι, καλά τα κοινωνικά προγράμματα, αλλά αν δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την ελευθερία, τότε προφανώς και κινδυνεύει η κοινωνική μας ευημερία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Αυστριακή και τη Ρουμανική Προεδρία. γιατί δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και ε, επέδειξαν ε, ιδιαίτερη τεχνογνωσία και όσοι φοβούνται το θέμα των σχέσεων με τον ΝΑΤΟ, να τους πω το εξής. Κοιτάξτε, στη δική μας την περιοχή ξέρουμε πολύ καλά τι είπατε. Είμαστε υπέρ αυτού του ταμείου, αλλά είμαστε και υπέρ του ότι το ΝΑΤΟ εγγυάται την ασφάλειά μας. Είναι ο εγγυητής της ασφάλειάς μας. Επ' αυτού δεν αλλάζει τίποτα και θα θέλαμε άλλες χώρες, η Γαλλία παραδείγματο χάρη, να δραστηριοποιηθεί για την προστασία της ε, ανατολικής πτέρυγας ε, του ΝΑΤΟ. Ε, Τέθηνε ερώτημα από τι ή πώς θα ωφεληθεί η Πολωνία. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι μπορούμε, αν συνεργαστούμε, να εξυγχρονίσουμε τον, τους εξοπλισμούς, τη βιομηχανία εξοπλισμών ε, και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης μπορούμε να προχωρήσουμε. Ελπίζω ε, τα κονδύλια αυτού του ταμείου να διατεθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάτι άλλο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να υπερψηφίσετε το κείμενο ε, όπως ακριβώς το διαπραγματευτήκαμε. Παρακαλώ να απορρίψετε όλες τις τροπολογίες υπέρ του 31CP και υπέρ όλων των τροπολογιών της Ολομέλειας, γιατί αλλιώς θα καταπέσει η συμφωνία μας. Αυτή είναι η θερμή μου παράκληση προς όλους σας. Ε, το γεγονός αυτό, όπως σας είπα, το έχω ενστερνιστεί, γιατί αποτελεί ευκαιρία για την αμυντική βιομηχανία, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ και για την βελτίωση των αμυντικών μας ικανοτήτων που είναι πολύ σημαντικές. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να επερασπιστούμε τον τρόπο ζωής μας και τον πολιτισμό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, συγχαίρω και ευχαριστώ τον ομιλητή. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Τώρα προχωράμε. Κοινή συζήτηση για τα καλυμμένα ομόλογα έκθεση του κυρίου Μπέρντ Λούκε και θα ακολουθήσει και μία άλλη συζήτηση για τα καλυμμένα ομόλογα και τα δημόσια εποπτεία. Είναι δύο εκθέσεις του κυρίου Λούκε. Κύριε Λούκε, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, για κάθε αγορά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ασφαλή, ασφαλείς κινητές αξίες. Γνωρίζουμε, δυστυχώς βέβαια, ότι αυτό σπανίζει. Γνωρίζουμε ότι οι τιτλοποιήσεις δεν προσφέρουν επαρκή κάλυψη. Αυτό το γνωρίζουμε το αργότερο από την χρηματοπιστωτική κρίση. Το γνωρίζουμε όλοι μας. Γνωρίζουμε επίσης ότι και τα κρατικά ομόλογα δεν προσφέρουν επαρκή προστασία. Ούτε και αυτά της Ευρωζώνης. Δεν δεν είναι ικανοποιητικά ασφαλή. Όπως σας είπα, το συνειδητοποίησαμε και με την κρίση του ευρώ και του δημόσιου χρέους. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν ε, τα καλυμμένα ομόλογα, ότι αυτά είναι ασφαλή τα καλυμμένα ομόλογα υπάρχουν εδώ και πάνω από 250 χρόνια και μέχρι τώρα ε, δεν έχουν καταρρέψει. Πρόκειται για μια κινητή αξία που την χρειαζόμαστε στην Ευρωζώνη και στην κεφαλαγορά. Γι' αυτό λοιπόν εκπλήσει το γεγονός ότι τα καλυμμένα ομόλογα δεν έχουν εξελιχθεί επαρκώς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι υπάρχει μόνο μία μικρή ομάδα κρατών που έχουν αυτή την παράδοση των καλυμμένων ομολόγων και την χρησιμοποιούν εδώ και πάρα πολύ καιρό, ενώ άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν σχεδόν καθόλου εμπειρία από καλυμμένα ομόλογα και δεν έχουν και σχεδόν καθόλου νομοθεσία για αυτά. Αυτό προσπαθούμε τώρα να αντιμετωπίσουμε εκδίδοντας ή ε, θεσπίζοντας, ψηφίζοντας οδηγία και κανονισμό για τα καλυμμένα ομόλογα. Η οδηγία είναι παράλληλα και το οδηγό νήμα για τις εξελισσόμενες αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που με τα καλυμμένα ομόλογα επιτυγχάνουν και αποκτούν ένα αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό εργαλείο. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, μπορούν να μεταφέρουν στην νομοθεσία τους αυτό που έχει αποδειχθεί σωστό εδώ και πολύ καιρό και που είναι μια πρακτική, δοκιμασμένη πρακτική στο θέμα των καλυμμένων ομολόγων. Όσον αφορά τη νομοθεσία, πραγματικά προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε στην πράξη όλα αυτά που αναφέρουμε, που πιστεύουμε για τις κινητές αξίες, όλα αυτά ε, για τα οποία διαπραγματευτήκαμε και νομίζω ότι τελικά καταλήξαμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Η οδηγία για τα καλυμμένα ομόλογα έχει τώρα λάβει τέτοια μορφή έτσι ώστε να έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες καλυμμένων ομολόγων. Αφενός εκείνα τα καλυμμένα ομόλογα τα οποία ορίζονται στον κανονισμό ε, περί επάρκειας κεφαλαίων, ομόλογα τα οποία προσέλκυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι είναι τα καλυμμένα ομόλογα υπό εξέλιξη, εκείνα που θα προσφέρουν νέες δυνατότητες χρηματοδότησης, θα εξετάσουν νέες δυνατότητες εξασφαλίσεων. Νομίζω ότι αυτές είναι πολύ καλές συνθήκες πλαίσιο, έτσι ώστε τα καλυμμένα ομόλογα να επικρατήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ικανοποιητικό χρηματοπιστωτικό εργαλείο και αυτές οι κινητές αξίες να γίνονται αποδεκτές και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε να θέσουμε πρότυπα σε διεθνές επίπεδο για αυτό το χρηματοπιστωτικό εργαλείο. Θα μπορέσουμε να τραβήξουμε την εμπιστοσύνη των ε, ε, πιστωτών και των ομολογιούχων. Ελπίζω όμως να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και το ενδιαφέρον των οντοτήτων, ε, των εκδότριων οντοτήτων, έτσι ώστε να ανοίξει η αγορά μας και να μην κλείσει έναντι εκείνων οι οποίοι επίσης ενδεχομένως ενδιαφέρονται για τη χρήση αυτού του εργαλείου. Νομίζω ότι κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Χαίρομαι για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει σήμερα Προσβλέπω στην αυριανή ψηφοφορία και βεβαίω θέλω να ελπίζω ότι αυτό το εργαλείο θα γίνει ευρέω αποδεκτό στην Κεφαλαϊκή Ένωση της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τώρα να δώσω το λόγο στην Επίτροπο Μπιερκόφσκα, παρακαλώ. μικρόφωνα παρακαλούμε. Τα καλυμμένα ομόλογα είναι μια σταθερή πηγή και αποτελεσματική προ το κόστο πηγή χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια τη κρίση. Ανταποκρίθηκαν καλά. Είναι πάρα πολύ δημοφιλή σε κάποια κράτη-μέλη, ενώ σε κάποια είναι κάτι καινούριο. Η πρόταση τη Κομισιόν προσπαθεί να αναπτύξει περαιτέρω αυτή την αγορά, βασιζόμενη στα υψηλά πρότυπα και τι καλέ πρακτικέ των εθνικών συστημάτων. Ε, πρόκειται για ε, ένα βασικό ε, στοιχείο τη αγορά κεφαλογορών. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πανευρωπαϊκή αγορά ομολόγων που θα υποστηρίζει το δανεισμό στην πραγματική οικονομία, χωρί να ενοχλεί ήδη τι εθνικέ αγορέ που λειτουργούν καλά θα υπάρξει όθηση της έκδοσης καλυμμένων ομολόγων στα κράτη-μέλη όπου είναι λιγότερο αναπτυγμένες αυτές οι αγορές. Οι κανόνες αυτές ε, θα σημαίνει ότι ε, θα υπάρχουν ασφαλή εργαλεία για τις τράπεζες που θα επιτρέψουν να χρηματοδοτήσουν τις εταιρείε και τα νοικοκυριά. Εκτιμούμε ότι η πιθανή εξοικονόμηση για τους δανειστές θα είναι περίπου 1,85 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επίσης, ε, θέλει η Ένωση να εναρμονίσει τους κανόνες προληπτικής εποπτείας προκειμένου να συνεισφέρει συνεισφέρουμε στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Το νέο πλαίσιο βασίζεται σε δύο πυλώνε. Καταρχήν σε μια οδηγία που παρέχει ένα κοινό ορισμό των καλυμμένων ομολόγων, παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των μέσων και εντοπίζει ε, τα περιουσιακά στοιχεία υψηλή ποιότητα που μπορούν να επιλεχθούν για να καλυφθούν από καλυμμένα ομόλογα. Επίση, έχουμε και την οδηγία για την εποπτεία ε, και θέτει του κανόνε για τις ε, ετικέτε. Και ο δεύτερο νομοθέτημα, ο ενισχύει του κανόνε για πρώτα μεταχείριση που θα, θα καλύπτουν τα ομόλογα που αγοράζονται από τράπεζε. Όπως ε, είδαμε στου τριμμέ διαλόγου και έχουμε και στη δήλωση της ε, Κομισιόν, η Κομισιόν θέλει να τροποποιήσει την ε, αναλογία για την κάλυψη ρευστότητα για να ρυθμίσει τα καλυμμένα ομόλογα. Αυτό θα, καλύψει, θα αντιμετωπίσει συγγνώμη, την επικάλυψη μεταξύ του ε, του αποθέματος ρευστότητας ε, αποθέματος αλλιές ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία. Ε, θα στείλουμε αυτά τα στοιχεία στο Κοινοβούλιο πριν από την ευριανή ψηφοφορία. Θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την επιτυχή για το επιτυχές αποτέλεσμα και κυρίως τον εισηγητή και όλους τους κοιόδες εισηγητές. Ο στόχος της πρότασης της Κομισιόν ε, διατηρούεται χάρη στην επικοδομητική προσέγγιση της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου και της καλή συνεργασίας με το Συμβούλιο. Η μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο και εφαρμογή των νέων κανόνων για τα καλυμμένα ονολογά θα πρέπει τώρα να προχωρήσει γρήγορα. Αυτό θα διασφαλίσει ότι έχουμε μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη προωθώντα τι ε, θέσεις εργασίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Επίτροπε, τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ροζάτη. Παρακαλώ, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εργαζόμαστε πάνω σε δύο έγγραφα, τα οποία ε, δημιουργούν νέες αρχές λειτουργίας για τα καλυμμένα ομόλογα. Πρόκειται για εγγυημένα ομόλογα και είναι ένα στοιχείο αυτό το οποίο δημιουργεί μια κεφαλιακή ένωση. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος που καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβιβασμό. Αυτά τα εγγυημένα ομόλογα ορίζονται δίνεται ορισμό του στο έγγραφο αυτό. Και τι είναι, είναι μια εγγύηση. Επίσης έχουμε δύο κατηγορίες εγγύσεων. Έχουμε τις ευρωπαϊκές που καλύπτουν τις προϋποθέσεις και έχουμε τις premium, οι οποίες επιπλέον καλύπτουν και τις απαιτήσει του κανονισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων, του CRR. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί από μόνη της να αποφασίσει για το πούλο του ενεργητικού και για το ρευστό. Καταλήξαμε σε ένα συμβασμό το 8% εγγύσεων για την ποιότητα των πιστώσεων. Επίσης υπάρχουν οι τραπεζικές εγγύσεις που γίνεται ένα έγγραφο υψηλής ποιότητας. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ τον βουλευτή, τον Ευρωβουλευτή Λούκε για την εξαιρετική αυτή έκθεση, αλλά επίσης και για την καλή συνεργασία που είχαμε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επικοδομητική της συμμετοχή. Ζητώ από όλους τους ευρωβουλευτές να υπερψηφίσουν χωρίς τροπολογίες αυτή την έκθεση. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Σαντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς για τα καλυμμένα ομόλογα, όπως ονομάζονται. Η διαδικασία ξεκίνησε εδώ το 2017 με μια έκθεση πρωτοβουλίας, η οποία θέσε και τις βάσεις του έργου μας για το νομοθετικό πακέτο που σήμερα έχουμε μπροστά μας. Δεν ήταν εύκολο, γιατί στην κάθε χώρα τα καλυμμένα ομόλογα έχουν εξελιχθεί διαφορετικά. Αποτελούν ένα χρηματοπιστωτικό εργαλείο, το οποίο έχει αποδείξει την αξία του κατά τους αιώνες έχουν βέβαια αναπτυχθεί διαφορετικά στις διάφορες εθνικές αγορές, αλλά έχουν νόημα. Και σε κάποιες αγορές όπως τη Δανία και τη Γερμανία τα καλυμμένα ομόλογα θεωρούνται ένα μέσο επενδυτικό πάρα πολύ συνηθισμένο. Σε άλλες χώρες όπως τη δικιά μου τη Μάλτα δεν υπάρχει καθόλου. Υπάρχει εδώ λοιπόν μια πολιτική πρόκληση μπροστά μας για να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο έτσι ώστε να προχωρήσουμε και στην ε, αγορά, ε, την, ε, μάλλον την ένωση της κεφαλαϊκής αγοράς. Ε, θα έπρεπε όμως να αποφασίζονται όλα από τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο ή θα έπρεπε να δεχτούμε τις διευθετήσεις που έχουν γίνει στις εθνικές αγορές μέχρι τώρα και που έχουν αποδείξει την αξία τους. Εγώ θα συμφωνούσα με το δεύτερο. Ε, δεν πρέπει να αλλάξουμε πράγματα τα οποία έχουν λειτουργήσει για δεκαετίες, για αιώνες ε, ικανοποιητικά. Βέβαια, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα μπορούσε να δημιουργηθεί με στόχο την προδευτική σύγκληση προς παρόμοιους κανόνες και πρακτικές. Το σεβαστικό κείμενο που έχουμε μπροστά μας ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτή την πρόκληση. Περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία της έκθεσης της Επιτροπής ΕΚΟΝ του 2018 και διορθώνει διάφορες πτυχές που θα ήταν μια ανησυχία για την ομάδα μου. Το κείμενο λοιπόν προωθεί την αναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενισχύει την διαφάνεια και την προστασία των επενδυτών, ενώ συγχρόνω αποφεύγει τον κίνδυνο ανατροπή των επιτυχημένων εθνικών συστημάτων καλυμμένων ομολόγων. Χαίρομαι που αυτέ οι προτεραιότητε αντικατοπτρίζονται στο κείμενο και κάνω έκκληση στο Σώμα να εγκρίνει αυτήν την πρόταση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα εκ μέρους του ΙΣΙΑΡ, ο κύριος Μαριάς, παρακαλώ. Πόση ώρα έχω κύριε Πρόεδρε. How much time I have, Mr. Chairman? Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. 30 seconds. Thank you. Και 30 δευτερόλεπτα. Στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη υπάρχει έντονος σκεπτικισμός για αυτού του είδους τα ομόλογα όταν φυσικά έχουν δει όλοι ότι ακόμη και κρατικά ομόλογα έχουν καταρρεύσει. Ιδίως στην πατρίδα μου όπου τα ελληνικά κρατικά ομόλογα τα οποία εμπιστεύτηκαν οι έλληνες πολίτες πάρα πολλοί μικρομεσαίοι συνταξιούχοι επένδυσαν ε, τους κόπους μιας ζωής στα ελληνικά ομόλογα και ήρθε μετά το περίφημο psi με απόφαση του eurogroup και κουρεύτηκαν τα ομόλογα αυτά κατά 53%. Και υπάρχουν σήμερα άνθρωποι στην Ελλάδα που είχαν εμπιστευτεί τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που δεν έχουν πλέον χρήματα να πληρώσουν τα φάρμακα να μπορέσουν να πάνε σε ένα νοσοκομείο. αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν έχουν καταρρεύσει τα κρατικά ομόλογα υπάρχει δυσπιστία απέναντι σε αυτή τη μορφή ομολόγου και φυσικά όπως αναφέρει στην εισήγησή του ο κύριος λούκε κάνει προσπάθεια η εισήγηση αλλά βεβαίως και ο κανονισμός να υπάρξουν οι μέγιστες εγγυήσεις ούτως ώστε αυτά τα ομόλογα να θεωρηθούν ασφαλή να έχουν φυσικά και πολλούς επενδυτές και έτσι να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως ένα εργαλείο το οποίο θα διαμορφώσει μια συνολική αγορά και ταυτόχρονα θα πάρει κοντά του και αρκετούς επενδυτές. όμως θα πρέπει να προσέξουμε πώς θα γίνουν αυτές οι διασφαλίσεις ούτως ώστε πραγματικά να μην φτάσουμε σε σημείο να καταρρεύσουν ακόμα και αυτά τα ομόλογα. όλα φυσικά κρίνονται από το πώς θα λειτουργήσει η αγορά. αν υπάρχει μεγάλη κρίση τότε πολλοί διερωτώνται αν και αυτά τα ομόλογα θα αντέξουν. ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Ναχτεγάλ τώρα. Η κυρία Ναχτεγάλ δεν είναι εδώ όμως. Οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκέρολτ. Ε, ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή που μπήκε μια ισορροπημένη και ρεαλιστική προσέγγιση. Η συμφωνία για τους κανόνες ε, σε ό,τι αφορά τα καλυμμένα ομόλογα εντάσσονται σε μια λογική που θέλει να ενισχύσει την Ένωση Κεφαλαγορών. Ε, είναι ουσιαστικό να μην ε, χάσουμε το στόχο, έσχατος σκοπός του νόμου που υθετούμε Στη συγκεκριμένη περίπτωση ουσιαστικά πρόκειται για την υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας. Βεβαίως προσπαθούμε να φέρουμε στις τράπεζες μια πηγή χρηματοδότησης ε, μακροπρόθεσμη για να ελοπιθεί ο στόχος αυτός. Τουλάχιστον θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να μην αποδυναμώσουμε το κανονιστικό πλαίσιο των τραπεζών. Καταρχήν, χωρίς αυτό να ε, σημαίνει ότι θα υπάρχει βελτίωση της χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις ε, και τους πολίτες. Και δεύτερον, αν αυτό ενέχει κινδύνους που ε, ουσιαστικά διακυβεύουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων είναι αξιοσημείωτο, γιατί θα επιτρέψει στις χώρες όπου δεν υπάρχουν ακόμη αγορές αυτές να ευνοήσουν τη δημιουργία ενός ε, εργαλείου ε, που ε, φαίνεται να είναι σταθερό ακόμη και σε περίοδους κρίσης και φέρθηκε ο συγητής. Άλλα εργαλεία όπως παραδείγματος χάρη μιας ευρωπαϊκής εγγύησης θα συζητηθούν περαιτέρω. Και καθώς τελευταία φορά παίρνω το λόγο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την καλή συνεργασία και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω να σας ευχηθώ. Καλό Πάσχα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια η κυρία Μπέρες. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το πλαίσιο της ελάχιστης εναρμόνισης των εθνικών καθεστώτων που θα δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι πρόσδεκτο. Θα μπορέσουμε να έχουμε ένα χρήσιμο εργαλείο επαναχρηματοδότησης και θα συνεισφέρει στην εμβάθυση των κεφαλαίων θα πρέπει να θυμηθούμε όμως ε, ότι ε, τα ομόλογα αυτά έχουν επιτρέψει στις τράπεζες να λειτουργήσουν σε δύσκολες συνδικές στην αγορά το 2008 παραδείγματος χάρη όταν είχαμε ε, το, το πόγιο της κρίσης. αυτά παίρνουν τα κύρια χαρακτηριστικά της κάθε εθνική αγοράς. Στη Γαλλία υπάρχει δυνατότητα να ε, έχουμε διαφορετικά στοιχεία κάλυψης. Ε, ε χάρη να έχουμε ε, και ε, δάνεια σε κίνητα αλλά και σε άλλες χώρες Δανία, Σουηδία, Ισπανία ε, και γι' αυτό έχουν εμπνευστεί από τις καλύτερες ε, πρακτικές με την δυνατότητα να έχουμε και αυτή την ευρωπαϊκή ετικέτα. Επίσης επιτρέπει στους πρωταγωνιστές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ετικέτα διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο και μπορούν να ευνοηθούν και οι επενδυτές ακόμη και σε περιόδους ε, που αντιμετωπίζουν προβλήματα οι τράπεζες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει κανένα το λόγο για το ΚΑΤΣΔΙΑΙ, έτσι λοιπόν θα δώσουμε το λόγο στην Επίτροπο για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας, για τις ε, παρεμβάσεις σας, ε, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία για αυτά τα καλυμμένα ομόλογα. Οι επενδυτέ εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζουν ότι αυτά τα χρηματοψηφιακά εργαλεία που αποκαλούνται ευρωπαϊκά καλυμμένα ομόλογα ή premium καλυμμένα ομόλογα, αυτά υπάγονται σε ειδική εποπτεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υπάρχει μια ισόρροπη προσέγγιση, να είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν οι βασικές διατάξεις. Ε, βεβαίως, εμείς θέλουμε να στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε τα καλυμμένα ομόλογα να γίνουν ακόμα πιο σημαντική πηγή χρηματοδότησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Πολύ ωραία, λέει ο πρόεδρο. Ε, τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, για άλλη μια φορά στον συνάδελφο κύριο Λούκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι, αγαπητοί στάλφοι. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδης ηγητές, κυρίως και τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολύ καλή συνεργασία κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής διαδικασίας. Νομίζω ότι τα σημαντικότερα ήδη ελέγχθησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Δύο μόνο παρατηρήσεις θα κάνω. Το πρώτο είναι ένα σύντομο σχόλιο ε, απευθυνόμενος προς τον κύριο Μαριά στον συνάδελφό μου. Βεβαίω και πρέπει κανεί πάντα να εξασφαλίζει ότι τα ομόλογα θα πληρώνονται πίσω. Παράδειγμα, τα κρατικά ελληνικά ομόλογα, παράδειγμα που μερικά δεν αποπληρώνονται. Εδώ όμω μιλάμε για άλλο πράγμα. Μιλάμε για ομόλογα τραπεζών. Άρα δηλαδή ε, υπάρχουν εξασφαλίσεις, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πουλ κάλυψης ε, το οποίο είναι προστατευμένο από παρεμβάσεις άλλων ομολογιούχων. Εγώ θα πρότεινα η ελληνική κυβέρνηση στο μέλλον να καταφύγει σε αυτή τη διαδικασία και τα κρατικά της ομόλογα να τα εξασφαλίζει μέσα από πραγματικές αξίες. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα καλό βήμα έτσι ώστε να βελτιωθεί και η αξιοπιστία της ελληνικής κυβέρνησης ως προς την δυνατότητα δανειοληψίας. Μετά, αυτά που είπε ο συνάδελφος ε, σχετικά ότι δεν είναι καλό να διαταράσει κανείς τις εύρυθμα λειτουργούσες αγορές. Ε, σωστό αυτό, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, γιατί αν δεν θέλει κανείς να διαταράξει καμία αγορά, ε, τότε θα πρέπει να επιτρέπει όλες τις πρακτικές και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιτρέπει και τις χειρότερες πρακτικές. Αυτό όμως δεν είναι ο στόχος της εναρμόνισης που επιδιώξαμε. Νομίζω τα καταφέραμε καλά να αποφύγουμε αυτόν, τον παραπλανητικό δρόμο. Με πώς με το να προβάλλουμε την ποιότητα της νομοθεσίας σε ορισμένα κράτη-μέλη. Και με τον τρόπο αυτό ασκούμε πίεση σε άλλα κράτη-μέλη να θελήσουν να προσαρμοστούν. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται γενικά η νομοθεσία για τα καλυμμένα ομόλογα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον τρόπο αυτό ανοίγουμε ένα πολύ καλό δρόμο για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η κοινή συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Συνεχίζουμε λοιπόν με το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξη ε, που είναι προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαπραγματεύσουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την νομοθετική πρόταση για το